Well, welcome to everybody. If you can sit, take your seat, please. We begin now. Παρακαλώ, καθίστε. Immediately. I will continue. Θα συνεχίσω στην Ιταλική. Αν φορέσετε τα ακουστικά σας θα είναι καλύτερα λέει. Πρόεδρος, σας καλωσορίζω. Καλωσορίζω τους φιλοξενούμενους μας, αλλά και τους συνάδελφους που είναι παρόντες εδώ σήμερα. Σήμερα το απόγευμα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία γι' αυτό που θα ονόμαζα μια στρατηγική γραμμή εργασίας τους επόμενους μήνες ως Επιτροπή Πολιτισμού. Και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με την παρούσα Προεδρία και με τη Λουξεμβουργιανή Προεδρία γιατί το θέμα αυτό έχει ευρύτατο ενδιαφέρον, δεν εξαντλείται στη σημερινή συγκυρία και θα ήθελα έτσι να έχουμε μια καλή εικόνα του τρόπου με τον οποίο θα συνεχίσουμε. Τα καινοτόμα σχολεία και η διδασκαλία στην ψηφιακή εποχή είναι ένα θέμα το οποίο προετοίμασε έτσι κι αλλιώς και η υπηρεσία τεκμηρίωσης per il lavoro fatto, eh, è stata una nostra proposta e ehm, Νομίζω ότι η πρότασή μας ε, έγινε δεκτή από όλες τις πολιτικές ομάδες, γιατί όπως σας είπα πρόκειται για ένα θέμα στρατηγικής φύσεως. Θα ξεκινήσω από μια γενικότερη σκέψη οι τεχνολογίες και το περιβάλλον, οι ψηφιακές τεχνολογίες και το ψηφιακό περιβάλλον συνιστούν μία επανάσταση στον τομέα της εκπαίδευσης και προκαλούν τεράστιες διαφορές στην διδασκαλία και τη μαθητεία και την δημιουργία επίσης της λεγόμενης δημιουργικής γνώσης, creative knowledge λέει στα αγγλικά η πρόεδρος. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές διδακτικού τύπου, παιδαγωγικού τύπου, σχολικού τύπου, νέες αίθουσες, νέες σχέσεις ε, ε, ανάμεσα στους ε, διδάσκοντες και στους διδασκομένους και θα πρέπει επίσης και να γνωρίζουν καλύτερα και να επηρεάζουν τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι διδάσκοντες έτσι ώστε οι αλλαγές να γίνουν και να γίνουν με την απαιτούμενη ταχύτητα. Ο κόσμος της σχολείου στην Ευρώπη δεν έχει αλλάξει και πάρα πολύ σε σχέση με την επανάσταση αυτή. Υπάρχουν αρκετά δεδομένα τα οποία θα το δείξουν αυτό. Το 75% των Ευρωπαίων φοιτητών και σπουδαστών διδάσκονται από δασκάλους και καθηγητές που δεν είναι ψηφιακά ενήμεροι. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των παιδιών γύρω στα 9-10 δεν έχουν τον εξοπλισμό για να διασφαλιστεί η πρόσβασή τους στο ψηφιακό κόσμο. Δεν υπάρχει υποδομή ε, για ψηφιακά βιβλία και το 75% των φοιτητών και μαθητών που έχουν κάποιες γνώσεις δεν έχουν επαρκείς και αποτελεσματικές γνώσεις. Ε, όλοι νομίζουμε ότι έχουμε προχωρήσει πολύ γρήγορα αλλά οι διαφορές είναι τεράστιες. Έχουν ανάγκη λοιπόν από υποστήριξη οι μαθητές και από το σχολείο και από τις οικογένειές τους και από τις πολιτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εμείς ακριβώς σαν πολιτικοί πρέπει να, να εντοπίσουμε τις στρατηγικές αυτές που θα βοηθήσουν να περάσουμε απέναντι από το ψηφιακό ρήγμα, να ενημερώσουμε σωστά τους εκπαιδευτές και τους διδάσκοντες, να προωθήσουμε την έρευνα, έτσι ώστε τα θέματα αυτά να μπορέσουν να προχωρήσουν. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τις νέες διαδικασίες εκμάθησης και πώς μπορεί να υποστηριχθούν από τα υπάρχοντα τεχνολογικά τρέντ, της τάσεις της τεχνολογικής και πώς θα εφαρμοστούν στα διάφορα επίπεδα παιδαγωγικής. Αυτά είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα. Υπάρχει ένα θέμα που αφορά ιδιαίτερα τους φοιτητές. Είναι η ιδιότητα του ψηφιακού σε εισαγωγικά πολίτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι μια προκλητική αν θέλετε ερώτηση η διαπίστωση ο λεγόμενος e-student, ηλεκτρονικός φοιτητής. Αυτό είχε τεθεί και στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ και η δυνατότητα χρήσης μιας ψηφιακής ηλικής κάρτας. Λοιπόν, είναι θέμα που αφορά και την τεχνολογία και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και τον ανταγωνισμό και την ε, μαθητική διαδικασία και ε, γενικότερα το ίδιο το περιεχόμενο ε, το, της διδακτέας ύλη. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους λοιπόν, να ευχαριστήσω τους δύο γενικούς διευθυντές τον Φιόλα και τον Μονέ, της DG Connect και της ε, DG Εκπαίδευσης, έτσι ώστε να μπορέσουμε και εμείς να βοηθήσουμε να υπάρξει μια συνέργεια ανάμεσα σε αυτές τις δύο σημαντικές γενικές διευθύνσεις και του αντίστοιχους επιτρόπους έτσι ώστε να υπάρξει ένας σωστός προσανατολισμός των τεχνολογιών των ψηφιακών και να υπάρξει και μια ουσιαστική ενίσχυση στις εκπαιδευτικές πολιτικές της Ευρώπης. Θα σας παρουσιάσω αμέσως τους ομιλητές, το πάνελ λοιπόν των εμπειρογνωμόνων μας. Ο πρώτος εμπειρογνώμων είναι η κυρία Κέρστι Λόγγ που έρχεται από το Ελσίνκι. Την ε, καλωσορίζουμε. Και μετά ο Βίνσεντ Τσόουντ από το Boston College, από τις Ηνωμένε Πολιτείες και την ευχαριστούμε για την παρουσία της. Έχουμε επίσης και το Γενικό Γραμματέα των Χριστών Δορυφορικών Πληροφοριών. Μαζί με τον καθηγητή Τσο έχουμε τον Ρόμπερ Χούμπνερ που είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή ε, της, ε, της εφαρμογές της τεχνολογίας της ψηφιακής από πλευράς της ΕΣΑ, της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας και τον εκπρόσωπο του Schoolnet που εκπροσωπεί 35.000 σχολεία στην Ευρώπη που θα μας δώσει μαρτυρίες λοιπόν δημιουργικού προγράμματος που ονομάζεται Classroom Lab, το εργαστήρι της τάξης. Εμείς γνωρίζουμε ότι ο χρόνος μας είναι σχετικά περιορισμένος, μια μισή ώρα περίπου, μια μισή ώρα, δυόμιση ώρες διορθώνει η πρόεδρος και γι' αυτό θα ξεκινήσουμε δίνοντας το λόγο στους δύο βασικούς εισηγητές, όχι πάνω από 15 λεπτά ο καθένας και στο τέλος των δύο ομιλιών τους θα υπάρξει ένας πρώτος γύρος ερωτήσεων και απαντήσεων και μετά θα δώσουμε το λόγο στους άλλους εισηγητές. Να προσθέσω σε μεθοδολογικό επίπεδο ότι πριν ξεκινήσουν οι ερωτοαπαντήσεις, εμείς τις τελευταίες αυτές ημέρες και με την υποστήριξη της DGCOM θελήσαμε να κάνουμε τη συνάντηση αυτή πραγματικά συμμετοχική και γι' αυτό συλλέξαμε και κάποιες ερωτήσεις από τα κοινωνικά δίκτυα. Ε, επιλέξαμε κάποιες από τις ερωτήσεις αυτές οι οποίες θα προσθεθούν στις ερωτήσεις των συναδέλφων. Λοιπόν, η καθηγήτρια ε, Σαλόνκα έχει το λόγο από την Φιλανδία. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Μεγάλη χαρά που βρίσκομαι εδώ και η τιμή. Ελπίζω να μπορέσω και εγώ να συμβάλλω σε μια κοινή ευρωπαϊκή κοινότητα προσπαθειών με αυτή την ε, σύντομη ομιλία. Καθήκον μου να μιλήσω για το ψηφιακό σχολείο για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν γνωρίζω πολλά, αλλά μπορώ να μιλήσω για τη Φινλανδία και ίσως θα μπορούσα να δώσω και μια ματιά ε, φουτουριστική, γιατί επιστημονικά στοιχεία μπορεί να μην έχουμε, αλλά έχουμε παρουσιάσει στην ε, μελέτη μας οράματα με βάση επιστημονικά στοιχεία και έρευνα. Έχω λοιπόν κάποια ζητήματα, ερωτήματα διατυπώ σε σχέση με τις ε, ε, δυνατότητες, ε, δεξιότητες για τον 21ο αιώνα. Και ένα σημαντικό θέμα το οποίο εμφανίστηκε πρώτο-πρώτο στα σχόλια σε σχέση με την εμπλοκή των σχολείων και τις ε, συναισθηματικές κοινωνικές δεξιότητες. Τι συμβαίνει δηλαδή στα παιδιά τα οποία θα κάθονται μπροστά σε έναν υπολογιστή, θα ασκούνται, θα κάνουν λιγότερη φυσική άσκηση κτλ. Άρα υπάρχουν αυτές οι ανησυχίες, αλλά ιδιαίτερα εμείς ε, στην Φιλανδία και θα δώσω και εγώ έμφαση στο παιχνίδι, στην, ε, στα τεχνικά, τη χειροτεχνία, τα χειροτεχνήματα και τη μουσική την αξιολόγηση που έχει πολύ μεγάλη σημασία φυσικά και στο τέλος θα σας δείξω και μια ταινία για κάτι το οποίο πολύ δύσκολα θα μπορούσα να περιγράψω με εποπτικά λοιπόν μέσα γιατί δεν θα μπορούσα να δώσω απάντηση στο πώς θα τα καταφέρουμε θα σας δείξω τι προτείνουμε. Το πρώτο λοιπόν ζήτημα δεν είναι τεχνολογία, είναι η μείωση της εμπλοκής του σχολείου, του engagement δηλαδή, που σε όλο τον κόσμο είναι φαινόμενο ορατό. Και το άλλο είναι το πώς μπορούμε να ζητήσουμε καινοτόμες νοοτροπίες εργασίας. Αυτό μπορείτε να το κοιτάξετε και στο περιβάλλον σας, τι είδους καινοτόμες μεθόδους ή νοοτροπίες εργασίας έχουν. Δεξιά βλέπετε παραδοσιακές μορφές εργασίας, αριστερά, ε, αριστερά βλέπετε παραδοσιακές μορφές εργασίας ε, και δεξιά τις καινοτόμες μορφές και Αν όμως αρχίσουμε μετά τα 12, τη 12 τον δεκαετή εκπαιδευτικό κύκλο να αναζητούμε τρόπο εμπλοκή σε καινοτόμε ε, συνθήκε εργασία θα είναι πολύ αργά. Θέλουμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε για του Ευρωπαίου πολίτε τη δυνατότητα προβλήματα περίπλοκα και μεγάλα να τα επιλύουν σε ε, ομάδα. Και άρα θέλουμε καινοτόμε ομάδε, θέλουμε ισχυρές ομάδες, θέλουμε πρακτική γνώσεως γιατί εγώ Φερρυπίν μπορεί να έχω μια γνώση σημαντική και να θέλω να την ε, στείλω μέσω του tweet σε όλο τον κόσμο, αλλά να μην έχω εδώ δυνατότητα επικοινωνίας με το διαδίκτυο και άρα δεν μπορώ να μεταδώσω την πληροφορία μου όπως θα ήθελα. Η εμπλοκή του σχολείου, όπως σας είπα, ριζικά μειώνεται. Η έρευνα του καθηγητή Σάρμιλαρς δείχνει ότι μπορεί η υπερκόπωση που μπορεί να εκδηλώνεται ήδη στο σχολείο ή να ξεκινάει στο σχολείο να εκδηλώνεται οριστικά και 20 χρόνια μετά. Άρα πρέπει να προσέξουμε πολύ εγκαίρως τις πρακτικές, τις συνθήκες στα σχολεία μας. Έτσι λοιπόν ε, ξεκινάμε ένα σχέδιο στην ε, Φιλανδία για το 2016, το οποίο δεν θα επεκταθεί σε ολόκληρη τη χώρα πάντοτε, αλλά σε συγκεκριμένα σχολεία θα δοκιμαστεί. Ε, θα κοιτάξουμε θέματα ε, τρόπου σκέψης, εκμάθησης, πολιτιστικές δεξιότητες, επικοινωνιακές δεξιότητες. Ξέρω ότι ε, έχουμε μόνο πολιτιστική προσέγγιση, τρόπο όμως και πολλαπλών δεξιοτήτων και γνώσεων, ικανότητες στους υπολογιστές του νούμερο 5 που είναι μετά από όλα τα προηγούμενα, γιατί πρώτα πρέπει να ξέρουμε τι ζητάμε και μετά το πώς θα το αναζητήσουμε και πώς θα το εγκαταστήσουμε. Και βέβαια δεξιότητες ε, συνδυασμού εργασίας και προσωπικού βίου και επιχειρηματικότητα. Αυτό για τις νέες ευκαιρίες και τη νέα οικονομική ε, ευημερία, το νέο οικονομικό πλούτο. Αυτό θα είναι κομμάτι του εθνικού προγράμματος σπουδών στη Φιλανδία. Έχουμε λοιπόν τη γενιά του Baby Boom, έχουμε τη γενιά X. Ξέρετε ότι και το ραδιόφωνο θα μείωνε την ανάγνωση. Η τηλεόραση θα καθιστούσε τον ε, τηλεθεατή παθητικό. Εγώ δεν θα έπρεπε να ήμουν εδώ δηλαδή σε θέση να σας κάνω ομιλία. Στην γενιά Y που ανήκει η κόρη μου γιατί γεννήθηκε το 1991, Ψηφιακή κάμερα, DVD και υπολογιστέ τα δεδομένα, αλλά η μικρότερη μου κόρη που γεννήθηκε το 1995 έχει γεννηθεί μέσα στην ψηφιακή ηλικία και δεν μαθαίνουν καν ε, το αλφάβητο με τη σειρά, ξεκινάνε με το όμικρο. Επίσης, ε, οι υποτιθέμενες πρακτικές και το λεγόμενο multitasking εγώ σα είπα ότι multitasking δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, πολλαπλή δηλαδή εκτέλεση εργασιών. Μπορεί κανεί να περνάει πολύ γρήγορα από τη μια λειτουργία στην άλλη, αλλά, το κάνει αλλά, κάνει, αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα να κάνει κανεί ταυτόχρονα πράγματα. Ωστόσο, τα παιδιά μπορούν και να εκτυπώνουν και να παρακολουθούν ψηφιακά και, να, και βέβαια έχουν πολύ μεγάλη εξάρτηση στα κινητά από τα κινητά μηχανήματα. Στο σχολείο όμως επί 7 ώρες δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Είναι σαν να βρίσκονται στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, να έχουν μπει δηλαδή σε ένα αεροπλάνο, να έχουν προσδεθεί και να περιμένουν να προσγειωθεί το αεροπλάνο για να ξανά έχουν επικοινωνία με τον υπόλοιπο κόσμο. Όλα αυτά τα στοιχεία της επικοινωνίας, της διαρκούς, της εντατικής μέσα από το διαδίκτυο το οποίο διαδίκτυο μετατρέπεται σε διαδίκτυο και αντικειμένων πλέον, αποτελούν την καθημερινότητα αυτών των παιδιών. Τώρα μιλούμε για κοινωνικοψηφιακές ε, συμμετοχές, ε, αναδιόμενες νέες αντιλήψεις, πρακτικές συμμετοχής κοινωνικής μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας. Και νομίζω ότι αυτό έχει σημασία όταν το δούμε σαν κοινωνικές πρακτικές και τρόπους επικοινωνίας. Αυτά λοιπόν κοιτάμε εμείς στη Φιλανδία. Κοιτούμε να δούμε αν υπάρχουν ε, Αν υπάρχει όντως αυτή η γενιά που έχει γεννηθεί μέσα στην ψηφιακή τεχνολογία, έχουμε αρκετά προηγμένες τεχνολογικές δυνατότητες, αλλά οι άνθρωποι αυτοί δεν ξέρουν καν ε, αν μπορούν να ξεβιδώσουν ένα κομπιούτερ ή να περιγράψουν τι έχει μέσα το μηχάνημα. Αυτή λοιπόν η ικανότητα χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας δεν σημαίνει και περίπλοκες τεχνικές δυνατότητες. Από τα παιδιά που ερευνήσαμε, 60% ήταν στη βασική χρήση, ε, ένα 30% ήταν στο παιχνίδι, χρήση για παιχνίδι και 10% μόνο είχε δημιουργική χρήση του υπολογιστή με παραγωγή είτε σε blogs είτε ε, ηλεκτρονικών παιχνιδιών από τα ίδια από μαθητές. Πρέπει να δούμε λοιπόν που βρίσκεται το κενό. Ποιος είναι ο μαθητής και ποιες ε, οι κοινωνικές ε, ικανότητες ή δεξιότητες μπορούν να έχουν καλύτερη απόδοση και επίδοση για το σχολείο. Φαίνεται να είναι θεωρητικό το ερώτημα Εκείνοι οι οποίοι φαίνεται ως μαθητές να έχουν περισσότερη κοινωνική δικτύωση, έχουν χειρότερες επιδόσεις ε, στα μαθηματικά, τα αγγλικά, τη γλώσσα, ε, εκείνοι, αυτοί που έχουν δημιουργική συμμετοχή στο χρήση των υπολογιστών, εκείνοι οι οποίοι έχουν ε, συμμετοχή ως προς τα παιχνίδια δείχνουν ακόμα χαμηλότερες επιδόσεις του σχολείο και ψηλότερο κινησμό από τους βασικούς χρήστες και αντίστοιχα κοιτούμε να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι από τους μαθητές οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν τη νέα αξία για την Ευρώπη. Το χάσμα λοιπόν, κοινωνικοψηφιακή συμμετοχή, η ευέλικτη χρήση των ε, ψηφιακών μέσων, το multitasking, ε, διάφορα εργαλεία της υπολογιστικής εποχής και αντίστροφα από την πλευρά του σχολείου και τις πρακτικές που τους προσφέρει. Έχουμε τα παραδοσιακά μέσα, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, γραφμικό ε, σύστημα, καθαρές διανοητικές δεξιότητες, χρήση του μολυβιού και του χαρτιού κτλ. Στην ε, προσήλωση που θα μπορούσαμε να καταγράψουμε. 50% καταγράφεται για τους ε, μέχρι 12 ετών Φινλανδούς, 4% δείχνουν άγχος, 5% κίνδυνο για ε, υπερκόπος, 15% κινησμό, 26% κίνδυνο κινησμού. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων κοινωνικο-συναισθηματικής νοημοσύνης και μάθησης είναι ένα περίπλοκο ζήτημα, αλλά προσπαθούμε να τους δείξουμε πώς μπορούν να αναγνωρίσουν, να περιγράψουν, να ε, ελέγξουν τα συναισθήματά τους μέσα σε μια κοινωνική και ψηφιακή συμμετοχή. Και επίσης αυτό που κάνουμε στην ψηφιακή ε, παιδεία στη Φιλανδία, αυτό είναι ένα περιβάλλον γνωστικό για τους δασκάλους για το μέλλον, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον το οποίο, στο οποίο μάλιστα συμμετέχουν ε, οι δάσκαλοι στο σύνολό τους σε εργαστήρια δημιουργικά δεν κάθεται δηλαδή κανείς πίσω από ένα κομπιούτερ, αλλά συμμετέχουν και με χειροτεχνική δουλειά ακόμη. 50% των νεαρών αποφύτων φαίνεται να έχουν προβλήματα στις ΗΠΑ ε, γιατί δεν έχουν μάθει τις σημαντικές κοινωνικές δεξιότητες που θα χρειαστούν στην περαιτέρω ζωή τους, όσο καλές γνώσεις και αν έχουν. Και η αξιολόγηση βέβαια, που έχει τεράστια σημασία, γιατί να έχουμε, για να έχουμε πραγματική γνώση θα πρέπει να έχουμε και γνήσια αξιολόγηση. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να αναπτύξουμε ένα σύστημα καθαρής αξιολόγησης στη Φιλανδία. που θα μπορεί έτσι να υποστηρίξει και τη γνήσια μάθηση, προσαρμογή δηλαδή των ε, μαθησιακών και κοινωνικών μοντέλων όπως έλεγα, έχουμε κάποιες καινοτόμες και πολλά υποσχόμενες πρακτικές. Έχουμε την μάθηση χάρη στην έρευνα, την διατύπωση προβλημάτων, την επίλυση πρακτικών περιστατικών ή φαινομένων. Εγώ ξέρετε από την ιατρική επιστήμη προέρχομαι, το έχω δει ήδη αυτό ανάγκη, ε, τη δυνατότητα για επεξεργασία ενός προβλήματος από τα παιδιά μέσα από το ίδιο το πρόβλημα που αποτελεί ένα τρόπο διδασκαλίας, μέσα από το παιχνίδι, μέσα από το παίγνιο και επίσης θα σας δείξω ένα βίντεο από την Βόρεια Φινλανδία, το Ούλου, που εάν με βοηθήσετε με τον σύνδεσμο ελπίζω ότι θα μπορέσω να σας δείξω. Γι' αυτό μάλιστα το βάζω στο τέλος πάντα, γιατί εάν δεν λειτουργήσει ο σύνδεσμος, διαλύεται όλη η παρουσίαση. Έχουμε λοιπόν αυτό το καινοτόμο σχολείο στη Βόρεια Φινλανδία. As an actor, I spend a lot of time oh, being someone else. Sorry. I was trying to skip it. This is how they study. They're very uh, architect, Heikki Luminen designed this school. It's an old school. because It was built 1983.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 θα ήθελα λοιπόν στο τέλος να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να απτυχθεί η κατάρτιση των διδασκάλων. Εδώ πρόκειται για μια πανεπιστημιακή σχολή κατάρτισης και βέβαια να συζητηθεί περισσότερο και να παρουσιαστεί ο τρόπος ανάληψης ηγεσία, παιδαγωγική βέβαια κατάρτιση, προσήλωση, ευημερία για τους νέους μας. Σας ευχαριστώ θερμά για το ενδιαφέρον σας. Very interesting presentation and I Σας ευχαριστώ πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση. Ασφαλώς θα ακούσουμε πολλά σχόλια και ερωτήσεις. Please. Καθηγητής Τσο. Βίνσεν Τσο από το Κολέγιο της Βοστόνης Θέλω να ευχαριστήσω τη συνάδελφο για το βίντεο, γιατί μου θυμίζει και γιατί ασχολούμαι με αυτή τη δουλειά. Μ' αρέσει πολύ να είμαι στο σχολείο και θέλω να είναι συναρπαστικό το σχολείο, να κάνει τη διαφορά και για μένα και φαντάζομαι ότι και για σας το ίδιο ισχύει. Στόχος μου είναι να δούμε λίγο τις προκλήσεις στο μέλλον, στην εκπαίδευση, αλλαγή της τεχνολογίας. Έχω κάποιες ιδέες να σας παρουσιάσω, χωρίς βέβαια να μπορώ να προτείνω λύσεις για όλα, αλλά νομίζω είναι ενδιαφέρον να σκεφτούμε και να συζητήσουμε. Έχω ένα ε, έγγραφο εκπονήσει και ασχολούμαι με τρία είδη τεχνολογίας και αυτό το σκελετό θα ακολουθήσω και στην παρουσίασή μου. Πρώτα απ' όλα όμως ε, ένα πείραμα σκέψης. Ας γυρίσουμε πίσω το 1991 όταν ε, η κόρη μου, η Generation Y όπως λέγεται, η γενιά Y γεννήθηκε, δηλαδή 24, 24 χρονών. Κάποιοι μπορεί να είστε σε αυτή τη γενιά ή να είχατε γεννήσει γύρω στα 91 τα παιδιά σας. Αυτό θα βλέπατε λοιπόν τότε έναν μεγάλο υπολογιστή που χρειάζεται για, αυτόν ένα floppy disk, μεγάλες κάμερες, ε, τηλέφωνα με καλώδιο, δεν μπορούσε κανείς δηλαδή να κυκλοφορεί στα δωμάτια και να τα χρησιμοποιεί τα ανασύρματα ή τα βιντεοσκόπια και μεγάλες βιντεοκασέτες. Καλό θα ήταν να δώσουμε ένα τέτοιο παλιό κομπιούτερ σε ένα παιδί και να δούμε τι θα πάθει όταν θα προσπαθήσει να τα χρησιμοποιήσει. Τι γίνεται λοιπόν είναι η ερώτηση όταν αλλάζει το σχολείο. Μπορώ να πάρω σήμερα ένα παιδί και να το βάλω πίσω στο 1991. Θα ξέρει το παιδί ε, πιστεύω όμω, πώ να κινηθεί, πώ να σταθεί με στην τάξη, τι να κάνει ακριβώ. Ψηφιακή επανάσταση. Αυτή η ιδέα ψηφιακή επανάσταση δεν είναι ε, μόνο μια ε, ερώτηση. Τρεις ερωτήσεις τουλάχιστον στο σύγγραμμά μου. Για τι είδους τεχνολογία, για το τι είδου αλλαγή μιλάμε για την τομέα πάντα τη εκπαίδευση. Έχουμε λοιπόν τρία επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο αφορά την επικοινωνία. Γνωρίζουμε ότι έχουμε την επιγραμμική μάθηση και το διαδίκτυο που οδηγούν σε νέους τρόπους μας. Δεύτερη αλλαγή, ε, ο εξοπλισμός, τα υλικά. Ε, τι βάζουμε στα χέρια των δασκάλων και των παιδιών. Κινητές, φορητές συσκευέ, υπολογιστές, Και τρίτο επίπεδο αλλαγής, το εκπαιδευτικό προσωπικό, δάσκαλος, ε, ο καθηγητής, τι γνωρίζει και τι μπορεί να δώσει στους φοιτητέ του για να του βοηθήσει ω υλικό. Αυτά λοιπόν είναι τα τρία επίπεδα αλλαγών, τα οποία σχετίζονται και με τρει διαφορετικού είδου τεχνολογίες εστίαση, focus technologies. Πρώτη είναι τα λεγόμενα, η λεγόμενη ανοιχτή ελεύθερη εκπαιδευτική πόρη. Δηλαδή βάζουμε τις πληροφορίες στο διαδίκτυο, εύκολη πρόσβαση, δωρεάν πρόσβαση για όλους. Ε, τα ηλεκτρονικά βιβλία κτλ. είναι ένα παράδειγμα ή βίντεο ή μαθήματα που γίνονται στο διαδικτύο. Όλοι μπορούν λοιπόν πολύ εύκολα να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις δυνατότητες μάθησης. Και όλα τα εμπόδια μπορεί κανείς να τα ξεπεράσει αν μπει στο διαδίκτυο και μπορεί να μάθει κάτι πάρα πολύ εύκολα οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Βασικά παραδείγματα είναι τα MOOCs ή ανοιχτά δηλαδή μαθήματα για όλους, ε, κάποια φόρουμ συζήτησης και η Ευρώπη έχει κάνει πολύ πρόοδο γιατί έχει καταστήσει προσβάσιμο τους σπόρους αυτούς, εφόσον είναι επιγραμμική online. Αυτό που θα ήθελα να σας θέσω ε, στη συζήτηση αυτή είναι και άλλοι τέτοιοι ε, εκπαιδευτικοί που Εδώ βλέπω ένα παράδειγμα, πώς σήμερα αντιμετωπίζει τη μάθηση ένας ε, φοιτητής. Πηγαίνει στο Twitter, ρωτάει στο διαδίκτυο online άλλους φοιτητές, ίσως μπορεί να καθοδηγηθεί μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Παράδειγμα, χάρη, σήμερα μπορεί κανεί να το κάνει αυτό για να βρει ένα καλό εστιατόριο, δεν το κάνει όμω για το σχολείο, στην εκπαίδευση. Ο λόγος για τον οποίο θέλω να προωθήσω τις τεχνολογίες αυτές είναι γιατί θέτουν το ε, ζήτημα να... αυτή η παραδοσιακή εκπαιδευτική πόρη, ε, η διδασκαλία είναι απαραίτητη ε, ή τι θα γίνει εάν χρειαστεί, ο, αν εξαρτηθεί πλέον ο φοιτητής και από τους ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους και θέλει συνέχεια να μπαίνει στο διαδίκτυο, κάθε μέρα και μόνο στο διαδίκτυο. Και μια άλλη ερώτηση. Πώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στη διδασκαλία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή τη τεχνολογία. Εγώ πρέπει να σα πω ότι προσπάθησα να παρακολουθήσω ένα online μάθημα. Όποτε έκανα λάθο σε μια ερώτηση, ένα quiz, άρχισα να απογοητεύομαι, τελικά εγκατέλειψα. Ε, διδακτορικό, αλλά πριν από λίγα χρόνια παρόλα αυτά έφυγα από ένα μάθημα, εγκατέλειψα. Μπορούμε να μιλήσουμε τόσο από αυτού του επιγραμμικού φοιτητέ για φοιτητέ ε, που έχουν ειδικέ ανάγκε που μπορεί να μην τα καταφέρνουν στην αίθουσα διδασκαλία. Αυτό σημαίνει το ίδιο θα του συμβεί και σε ένα online μάθημα. Μπορεί να χρειάζεται, παραδείγματο χάρη, ένα ε, τυφλό σε ένα ειδικό σύστημα για να ακούει. Ε, ο κουφό μπορεί να χρειάζεται ένα διερμηνέα τη νοηματική κτλ. Έχουμε λοιπόν αυτό το θέμα των υλικών, του εξοπλισμού που βάζουμε στα χέρια των ε, φοιτητών και των ε, δασκάλων. Ακούσατε και για το net computing και πρέπει να έχει πρόσβαση ο μαθητής σε υπολογιστή, σε μια ταμπλέτα, όλη τη μέρα, για όλα τα μαθήματα. Ελπίζουμε ότι αν υπάρχει πρόσβαση στο σχολείο σε περισσότερη τεχνολογία θα δούμε και να αναδύονται νέες μορφές και μάθησης δηλαδή μπορεί να μπαίνουν στο διαδίκτυο οι μαθητές και να αναζητούν πληροφορίες για ένα θέμα, να δημιουργούν ένα project, να βρουν κάποια βίντεο, να ενημερώνουν το κοινό, δημοσιεύοντας αυτά τα οποία έμαθαν κτλ. Και έτσι βλέπουμε μια επανάσταση στον τρόπο δασκαλίας. Αυτό βέβαια δεν συμβαίνει παντού, αλλά η ελπίδα μας αυτή είναι. Σε ό,τι αφορά τώρα την έγκριση αυτών των προγραμμάτων, είμαστε στην Ευρώπη ηγέτες, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε τέτοιο εξοπλισμό. Στην Νότια Αμερική έχουμε την Αργεντινή που έχει εταιρικέ σχέσει με την εταιρεία Intel και είχαν πάρα πολύ καλά νούμερα και στη χώρα αυτή. Ε, υπάρχουν βέβαια και κάποιοι περιορισμοί και κάποιε επιφυλάξει. Σίγουρα είναι περιορισμένοι ε, ε, τοπικά αυτοί οι πόροι, αυτές οι συσκευές και δεν σημαίνει ότι πολύ απλά και μόνο η διάθεση αυτών των, η κατοχή αυτών των συσκευών βοηθά να διδάξεις καλά. Υπάρχουν καταστήματα της ανάπτυξης ε, των παιδιών. Μπορεί να μην ε, ωφελούνται και τόσο πολύ τα παιδιά από το να έχουν τόσο ε, μεγάλη πρόσβαση σε τόσες πολλές πληροφορίες, τόσο εύκολα, γιατί μπορεί να είναι σε βάρος άλλων καταστάσεων, του να έχουν μια συναισθηματική κατανόηση και εκπαίδευση κτλ. Επίσης μια άλλη ιδέα είναι η λεγόμενη ψηφιακή ηθαγένεια. Έχουμε γεννηθεί ε, στην ε, τεχνολογία τη ψηφιακή, αλλά δεν έχουμε μάθει να την διαχειριζόμαστε με ηθικό τρόπο και υπεύθυνο τρόπο και να λαμβάνουμε πάντοτε τις πιο σωστές αποφάσεις για τη χρήση της τεχνολογίας. Τρίτο επίπεδο αλλαγής, είπα, είναι ο καθηγητής, ο δάσκαλος, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε το δάσκαλο να διδάξει το μαθητή. Έχουμε τα συστήματα δεδομένων υπολογιστή. Έτσι έχουν καλύτερα πληροφορίε στη διάθεσή τους οι δάσκαλοι για να καλύψουν τα κενά. Ε, αν ξέρουν τι θέλουν να μάθουν και τι πρέπει να μάθουν οι μαθητές, μπορούν να διδάξουν καλύτερα οι δάσκαλοι. Ε, παλιά, τον παλιό καιρό που εγώ ήμουνα θητητής, έτσι μάθαινα. Πήγαινα δηλαδή σε ένα γραφείο, έμενα ώρες ολόκληρες, ανοίγοντα σιρτάρια, κλείνοντα σιρτάρια και ίσως να μάθαινα και κάτι για τα παιδιά. Σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να αξιολογούμε τους μαθητές, να συλλέγουμε πολλές πληροφορίες ε, κάποιες μπορούν να αφορούν ε, θεωρητικές, ε, κοινωνικές επιστήμες, δοπισκές επιστήμες κτλ. Μπορούμε όμως να συλλέξουμε και στοιχεία για την εργόμενη συναισθηματική ε, νοημοσύνη και για το αν το παιδί νιώθει χαρά, ικανοποίηση στο σχολείο, αν νομίζει ότι κάνει πιο δίκαιο τον κόσμο κτλ. Όλα αυτά μπορείτε τα βάλετε στο κομπιούτερ. Και έτσι παίρνουν ένα feedback οι δάσκαλοι για το πώς εξελίσσεται τα πράγματα. Τι μαθαίνουν ε, τι πρέπει να μάθουν την επόμενη εβδομάδα, τον επόμενο μήνα, πώς πρέπει να παρέμβω για να προοδεύσουν όλοι μου οι μαθητές και ούτω καθεξής. Και όπως γνωρίζετε επίσης υπάρχουν και πολύ μεγάλες παραλλαγές και ε, διαφοροποιήσεις για το πώς μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει ανάλογα με το κράτος μέλος ε, τα διάφορα στοιχεία έχουμε διαφορετικά συστήματα λογοδοσία ή διαφορετικούς λόγους για τη χρήση κάποιων δεδομένων. Στον τομέα της τεχνολογίας επίσης, υπάρχει το πρόβλημα της πρόσβαση. Ποιο έχει πρόσβαση σε ποια δεδομένα σε άλλους ε, τόπους, σε άλλα μέρη μπορεί οι δάσκαλοι να έχουν πρόσβαση διαφορετικά δεδομένα. Άρα τι γίνεται, ακολουθούν τα δεδομένα το μαθητή, αν περάσει από το ένα σχολείο στο άλλο. Μήπως πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή ο ε, καθηγητής. Ή καλό θα ήταν να μελετήσει τα στοιχεία που έδινε το προηγούμενο σχολείο και να μπορέσει πάνω από εκεί να ε, βασιστεί. Τώρα, στήριξη αυτή τη χρήση τεχνολογία. Ε, σίγουρα πρέπει να συμβούν κάποιε διαθροτικέ αλλαγέ, δηλαδή εκπαίδευση των εκπαιδευτών, να έχουν το χρόνο για τη χρήση και των υπολιστών ε, των στοιχείων αυτών και συζήτηση με τα παιδιά. Τι λειτουργεί για αυτά, τι δεν λειτουργεί, τι μπορεί να γίνει. Και επίση βελτίωση τη ροή δεδομένων και πώ μπορούν να συνομιλούν μεταξύ του οι μαθητέ και οι φοιτητέ. Υπάρχει επίση και ένα ευρύτερο ζήτημα, το οποίο έχει να κάνει με το όλα πρέπει να ε, έχουν να κάνουν με την παραδοσιακή ακαδημαϊκή μάθηση. Τι είναι εκπαίδευση τελικά. Είναι πολύ καλή η χρονική στιγμή να σκεφτούμε οι αυριανοί ενήλικοι, τα παιδιά πώς θέλουμε να εξελιχθούν. Τι κοινωνικές δεξιότητες θέλουμε να έχουν ε, αναπτύξει. Και βέβαια να έχεις μια ιδέα για το πώς θέλει να εξελιχθούν τα παιδιά, μπορείς να συλλέξεις τα σχετικά δεδομένα. Μίλησα λοιπόν για τις τεχνολογίες, για τις προκλήσεις, για κάποιες ευκαιρίες και δυνατότητες και τώρα έχω κάποιες γενικές ε, σκέψεις που θα ήθελα να αναφέρω. Πρώτα απ' όλα, σίγουρα είναι καταπληκτικό που έχουμε τόση τεχνολογία σήμερα. Αλλά τελικά δεν μιλάμε για τεχνολογία, αλλά για ανθρώπου. Τεχνολογία είναι το εύκολο κομμάτι. Οι άνθρωποι, ο άνθρωπο είναι η πρόκληση να πιστέψει, να καταλάβει, να θέλει να χρησιμοποιήσει αυτές τις τεχνολογίες όπου είναι διαθέσιμες και όπου μπορεί να τις χρησιμοποιήσει. Το δεύτερο θέμα είναι ότι ναι μεν βλέπουμε αύξηση της χρήσης των διαφόρων μέσων, online, στις αίθουσες δασκαλίες, πληροφορίες που συλλέγουν οι δάσκαλοι κτλ. Πρέπει όμως να παραμείνουμε διαδραστικοί, να δούμε δηλαδή προβληματίζονται από κοινού, έρχονται από κοινού οι άνθρωποι, πειραματίζονται με νέε ιδέε. Γιατί αυτό που θέλουμε ουσιαστικά να προωθήσουμε είναι την κοινωνική αλληλεπίδραση, γιατί έτσι μαθαίνουμε. Και το τρίτο ερώτημα είναι τι παραμένει ίδιο. Με άλλα λόγια, με τεχνολογία έχει βελτιωθεί η ζωή μας. Με το email βελτιώθηκε η ζωή μας. Τόσο πια. Ίσως το 91 εκεί στις παλιές αίθουσες δασκαλής είναι κάτι που θα πρέπει να μας απασχολήσει και να δούμε τι γινόταν τότε. Γιατί μπορεί με τεχνολογία να μην μπορεί να γίνουν κάποια πράγματα, εξακολουθούν όμω να είναι πολύ ωραία αυτά τα πράγματα και ίσως πρέπει να τα σκεφτούμε. Στην όλη πορεία τη ανθρώπινη ανάπτυξη, αυτή η ψηφιακή επανάσταση που έχουμε σήμερα είναι ε, μόνο ένα ε, στοιχείο. Δείτε όλα αυτά. Ε, έχω και τις, ε, τα στοιχεία μου. Βλέπετε το ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο και τη διεύθυνσή μου στο Twitter. Πρώτα σε επαφή. Ευχαριστώ. Thank you. Thank you so much. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τους δύο μιλητές για τις σκέψεις τους πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Σε αυτή τη φάση τώρα θα ήθελα να ξεκινήσω την δυνατότητα να τεθούν ερωτήσεις από συναδέλφους και να δοθούν απαντήσεις πριν περάσουμε στο δεύτερο πάνελ. Πρώτα όμως θα ήθελα να φέρουμε στην επικαιρότητα, στην επιφάνεια τις ερωτήσεις αυτών οι οποίοι μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα ενδιαφέρθηκαν. Η πρόεδρος του European Youth Forum είναι η πρώτη, δεν μπορούσε να είναι παρούσα. Έχουν ένα συγκεκριμένο ερώτημα όμως, το οποίο συνθέσαμε κατά κάποιο τρόπο. Θα μπορέσουν οι δύο μιλητές να απαντήσουν, ίσως και οι επόμενοι. Τη διαβάσατε ελπίζω την πρώτη ερώτηση. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν, υπάρχει ένα πρόβλημα. η πρώτη έλεγε μπορούν οι να ενταχθούν στις διδακτικές διαδικασίες. Η δεύτερη από τον κύριο Φρίκε ή την κυρία Φρίκε μάλλον Λοιπόν, πώς μπορεί κανείς να δει τα θέματα αυτά με πιο συνολικό, ολιστικό σχεδόν τρόπο και να εντάξει τις τεχνολογίες αυτές λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές επιπτώσεις στη μαθησιακή διαδικασία και πώς μπορεί να κινητοποιήσει την αίσθηση υπευθυνοποίησης μέσα από τη χρήση των τεχνολογιών. Κοινωνική ευθύνη μέσω της τεχνολογικής καινοτομίας. Εδώ μιλάμε για το digital divide, το ψηφιακό ρήγμα. Και υπάρχει και μία συγκεκριμένη ερώτηση σε σχέση με αυτό. Εάν πράγματι το ρήγμα αυτό μπορεί να καλυφθεί μέσα από την εκπαίδευση ή και μέσα από την παροχή ειδικών πολιτικών που να βοηθήσουν τα παιδιά να λειτουργούν όχι μόνο ανταγωνιστικά στον τομέα των σχολικών. Λοιπόν, αυτές ήσαν οι ερωτήσεις. Συγκεντρώνουν αρκετές ε, περισσότερες ερωτήσεις. Ε, δεν θα ε, μείνω εδώ για να μπορέσετε να απαντήσετε, αλλά θα δώσω πρώτα το λόγο στους συναδέλφους. Ο συνάδελφος Σδροζεύσκη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους δύο ομιλητές για τις πληροφορίες τις οποίες μας έδωσαν. Έχω κάποιες ερωτήσεις που συνδέονται κυρίως με μια τάση την οποία διαπιστώνουμε. Εδώ και 100 χρόνια η Ευρώπη είχε σαν στόχο να πάνε όλα τα παιδιά στο σχολείο. Η επόμενη φάση ήταν να αυξηθεί η υποχρεωτική σχολική περίοδος και το επόμενο βήμα ήταν ο εκδημοκρατισμός των σχολείων και η δημιουργία σχολικών συμβουλίων με παιδιά και γονείς. Και τώρα είναι η τεχνολογία η οποία θα πρέπει να μπει σε όλα τα σχολεία στην Ευρώπη. Κατά κάποιο τρόπο έχω την αίσθηση ότι κινδυνεύουμε να πέσουμε σε μία παγίδα, δηλαδή ε, απομονώνουμε κάποια από τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και αυτά αντιμετωπίζουμε. Σε πολλά σχολικά συμβούλια οι γονείς και οι δαιμόνες έχουν ξεπεράσει τα αιτήματά τους, έχουν λειτουργήσει ε, εκτός λογικής μερικές φορές. Να πω επίσης ότι πάρα πολλοί καθηγητές, όχι όλοι αλλά πάρα πολλοί δάσκαλοι και καθηγητές δεν παρακολουθούν την τεχνολογία και την ταχύτητα με την οποία αλλάζει η τεχνολογία. Τρίτον, υπάρχουν κάποια πρώτα βήματα ενιοποίησης ε, της διδασκαλίας, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα σχολεία. Και αυτό δεν ισχύει μόνο στο εσωτερικό της Ευρώπης, αλλά και σε όλον τον κόσμο έχουμε να αντιμετωπίζουμε διαφορετικά θέματα, διαφορετικές συγκυρίες και η τεχνολογία από μόνη της δεν αρκεί. Προφανώς και εγώ χρησιμοποιώ το διαδίκτυο για εκπαιδευτικούς λόγους, αλλά βλέπω στο περιεχόμενο του διαδικτύου πάρα πολλά λάθη σε ονόματα, σε ημερομηνίες, σε ερμηνείες. Το μέγεθος, ο όγκος αυτών των λαθών στην ουσία αυτοεξυπηρετείται και αυξάνεται συνεχώς. Το να θεωρήσει κανείς ότι το διαδίκτυο ε, είναι ένα κατεξοχήν εκπαιδευτικό μέσο είναι παραπλανητικό. Είπα βέβαια στην αρχή ότι η εκπαίδευση πέφτει μέσα σε μια παγίδα σε σχέση με την τεχνολογία και εδώ έρχεται αυτό το 10% της δημιουργικότητας που απαιτείται και στην οποία αναφερθήκατε. Το ποσοστό αυτό θα πρέπει να αυξηθεί. Τα παιδιά σαν παράδειγμα παίζουν παιχνίδια online. Αν αυτό δημιουργεί στρες, κινησμό και τελικά έλλειψη δημιουργικότητας, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει και να βγάλουμε τα κατάλληλα συμπεράσματα. Οι αναλύσεις λοιπόν τις οποίες έχετε κάνει δείχνουν αρνητικές συνέπειες ψυχολογικές, κοινωνικές ή οτιδήποτε άλλο. Ευχαριστώ συνάδελφε. Ε, πραγματικά ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και πυκνή η ερώτησή σας, αλλά να είσαστε σύντομοι γιατί έχουμε άλλες πέντε σημαντικές εκθέσεις. Ντιμπάτσκα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα ξεκινώντας να εκφράσω μια σκέψη. εκείνοι οι οποίοι διερωτώνται πού πήγε όλη αυτή η σοφία. Θα πω το εξή. Τη σοφία την έχει δικαταστήσει η διδασκαλία. Τη διδασκαλία δε η πληροφορία. Να θυμάμαστε λοιπόν το εξή. Ότι είναι μεγάλο το πλεονέκτημα να έχουμε ευχερή πρόσβαση στην πληροφορία. Αλλά υπάρχει και ένας μεγάλος κίνδυνος να γίνει πιο ρηχή η πληροφορία. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν χρησιμοποιούμε τα ηλεκτρονικά μέσα, την ηλεκτρονική τεχνολογία, να διατηρούμε και την διαπροσωπική σχέση. Τη σχέση μεταξύ δασκάλου και μαθητή, για να διατηρείται αυτή η προοπτική. Γιατί αν κινδυνεύσει η διαπροσωπική, ανθρώπινη σχέση, εάν περάσουμε σε έναν ψηφιακό κόσμο, ο οποίος θα αντικαθιστά ως εικονικός κόσμος τον αληθινό, τότε πολύ φοβούμαι ότι η γενιά θα πάρει το όνομα διαλυμένη γενιά. Πρέπει βεβαίως να παρακολουθήσουμε τη τεχνολογία, αλλά με σωστή πρόπτικη. Και θα απαντήσω στον συναδελφό Στραγεύσκη πως λυπούμε που δεν έχει ρίξει μια ματιά στην έκθεσή μου συνάδελφος για την έκθεση της Πολόνια όπου λέω ότι ναι υπάρχει συνεργασία αλλά συνεργασία μέσα από τη διαφορά. Η διαφορά είναι ο λόγος της υπερηφάνειας που αισθανόμαστε ως Ευρωπαίοι. Δεν σημαίνει πρέπει να την διαλύσουμε. Σύντομα μόνο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ο ρόλος του σχολείου στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων δεν είναι τόσο σημαντικός όσο πιστεύουμε μερικές φορές. Το μικρό παιδί, ακόμα και το πολύ μικρό, αποκτά δεξιότητες μέσα στην οικογένειά του ή στην διαπροσωπική επαφή με τους φίλους του. Καλό είναι όμως να ανοίγουν τα θέματα αυτά για συζήτηση. Και θυμούμε στην αρχή της δεκαετίας του 90 όταν είχε αρχίσει η αργή επέκταση του ψηφιακού κόσμου, όπου θέλαμε όσο δυνατόν περισσότερο να έχουμε την επαφή μέσω των τεχνολογιών. Στη δεκαετία που ακολούθησε επιδιώκαμε τη βέλτιστη δυνατή χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, στην καθημερινή μας ζωή, στη μάθηση, στο χώρο εργασίας. Ενώ τώρα, αυτή τη δεκαετία, αρχίσουμε να εκφράσουμε τους φόβους για το τι είδους κινδύνους μπορεί να συνεπιφέρει αυτή η ψηφιακή τεχνολογία και κυρίως για τα μικρά παιδιά. Όλοι τον ίδιο φόβο εκφράζουμε. Το φόβο ότι τα παιδιά θα αρχίσουν να απολένουν την κοινωνική τους ευθύνη, τις, κοινωνικές δεξιότητες, επειδή αποκτούν τις ψηφιακές δεξιότητες. Ερωτώ λοιπόν, υπάρχει κάποια μελέτη που να καλύπτει το πρόβλημα αυτό και για άλλη μια φορά ευχαριστώ τους δύο προσκεκριμένους για τις εξαιρετικές παρουσίες. Ευχαριστώ κύριε Γόρνου. το λόγο. Uh, thank you. I find... Σας ευχαριστώ. Είδα ότι και οι δύο αυτές ε, παρεμβάσεις ήσαν εμπνευσμένες. Μοιάζουν αυτά τα οποία έκανα πριν ασχοληθώ με την πολιτική και είναι πολύ ενδιαφέρον να βλέπει κανείς τέτοιου είδους ε, παρεμβάσεις was Sugata Mitra who developed um, uh, Ο συνάλφος Μίτσελ είχε ασχοληθεί με τα θέματα της ε, ε, εκμάθησης μέσω της χρήσης ε, της πληροφορικής και γενικά η ψηφιακή γνώση και η διαδικτυακή γνώση και διδασκαλία δεν πρέπει να περιορίζονται σε ένα κομπιούτερ. Ε, είδαμε ότι τα παιδιά τώρα πια δεν χρειάζεται να μάθουν απλά να μιλήσουν ή να περπατήσουν, αλλά και να ασχοληθούν με θέματα πληροφορικής και ιδιαίτερα τα παιδιά με ειδικέ ανάγκες, εκεί έχουν ε, πολλές δυνατότητες. Ε, τώρα, για το τι χρειάζεται η ψηφιακή εκπαίδευση, αυτό είναι, στόχος είναι να δημιουργήσει νέους ανθρώπους φιλοπερίεργους, με διερευνητικό πνεύμα οι οποίοι θα γίνουν ενεργοί πολίτες στο μέλλον. Γενικά η πολυγλωσία σε, στα σχολεία, η επαφή με τη φύση, η, φυσικά η ψηφιακή εκπαίδευση, η χειροτεχνία, όλα αυτά βοηθούν. Ε, βέβαια πρέπει να καλύψουμε και τις ανάγκες των παιδιών πριν φτάσουμε σε αυτό. Αν τα παιδιά πεινάνε, είναι δυστυχή, οι οικογενειακές τους ζωές είναι δύσκολες, προφανώς το σχολείο δεν θα βοηθήσει. Πρέπει όμως το σχολείο να δώσει ευκαιρίες και οι ευκαιρίες αυτές υπάρχουν. Ε, δεν θέλω να φανεί ότι κηρύττω εδώ με αυτά τα οποία λέγω, αλλά εν πάση περιπτώσει θέσω μια ερώτηση. Ε, οι καθηγητές των παιδιών μου είπαν ότι βασικός τους στόχος είναι να διασφαλίσουν την ευτυχία των παιδιών, γιατί αν είναι ευτυχή τα παιδιά τότε μαθαίνουν και θα πρέπει να δούμε ε, τις εικόνες που είδαμε, πού νιώθουν άνετα τα παιδιά, όχι όταν είναι σε θρανείο βέβαια, όχι όταν συνειδητοποιούν ότι αξιολογούνται και εξετάζονται, αλλά όταν είναι αυθόρμητα δημιουργικά τα παιδιά, ανεξαρτήτως του τελικού αποτελέσματος, η διαδικασία μετράει. Ανησυχώ λοιπόν για τον τρόπο με τον οποίο επανέρχονται ορισμένες χώρες σε βικτοριανές αρχές σχολικής αυστηρότητας και όχι ε, μαθητικής ε, ε, δραστηριότητας και τα παιδιά στρεσάρονται, πιέζονται και δεν προετοιμάζονται για τον κόσμο τον οποίο ζούμε. Λοιπόν, ε, θα πρέπει αυτά τα ιδιαίτερα δίσκαμπτα πλαίσια, πιεστικά πλαίσια να τα ε, ελαφρύνουμε. Τρούπελ. Ακούσαμε τρεις ομιλητές και σίγουρα υπάρχουν ε, κάποιες αρνητικές επιπτώσεις ε, με τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών. Στο σχολείο εγώ όμως θέλω να εστιάσω ε, στις ικανότητες των δασκάλων. Λέτε ότι αν δεν είναι προσιλωμένα τα παιδιά στο σχολείο μπορεί και να μην ενδιαφέρονται να μάθουν. Ε, γιατί βλέπουν και ότι ο δάσκαλος έχει μείνει πίσω. Άρα σήμερα τι αιτήματα έχουμε από τους δασκάλους, τι απαιτήσει έχουμε από αυτούς, γιατί πράγματι πρέπει να ξέρουν να έχουν ψηφιακές δεξιότητες για να μπορέσουν ε, να έρθουν σε επαφή με τους ε, μαθητές τους, αλλιώς δεν υπάρχει πραγματική επαφή, να γνωρίζουν πολλά λοιπόν για τις ψηφιακές συσκευές. Από την άλλη πλευρά όμως, Υπάρχει και μια προσέγγιση εξίσου μοντέρνα, θα τη χαρακτήριζα και παραδοσιακή, ότι δηλαδή οι δάσκαλοι πρέπει να μπορούν να δίνουν προσανατολισμό, καθοδήγηση, υποστήριξη και θα μπορούν να δείχνουν ότι μπορούν να διαχειριστούν την ψηφιακή ε, χρήση, το ψηφιακό περιεχόμενο. Εσείς έχετε κάποια πορίσματα και αν ναι, ποια είναι αυτά και αν έχετε κάποιες ανησυχίες για τις ε, δυνατότητες, ικανότητες, ε, δεξιότητες των εκπαιδευτικών. Λουίτζι Μόργαν ο τελευταίος. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω τους ομιλητές και για τις προτάσεις τους μεταξύ άλλων. Νομίζω ότι υπάρχουν δύο πτυχές που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Να ε, είναι οι μαθητές και αφετέρου είναι οι εκπαιδευτικοί. Δεν υπάρχει αμφιβολία ως προς το ότι το πραγματικό πρόβλημα σήμερα για τα μικρά παιδιά. Ε, είναι διαφορετική κατάσταση στο σχολείο, στο δημοτικό, σε σχέση με το πανεπιστήμιο, για παράδειγμα. Η κάθε γενιά μαθαίνει με διαφορετικό τρόπο. Και δεν είναι μόνο η τεχνολογία το θέμα. Σίγουρα βέβαια και με την πρώτη τεχνολογία αλλάζει και ο τρόπος εκμάθησης. Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε βέβαια στην τεχνολογία της συγκεκριμένη χρονική τύπης κάθε φορά δεν θα ήταν αυτό παραγωγικό. Σημαντικό είναι να έχουμε υπόψη μας και την κοινωνική και συναισθηματική νοημοσύνη. Γιατί δεν αρκεί να μαθαίνει κανείς συγκεκριμένα πράγματα. Αυτή η τεχνολογία μπορεί να δώσει απαντήσεις, Τι θέλω να πω με όλα αυτά. Είναι σημαντικό να συζητούμε για το σχολείο. Σίγουρα πρέπει να δούμε πώς αξιοποιείται η νέα τεχνολογία στη διδασκαλία, αλλά υπάρχουν και άλλες πτυχές. Οι γνώσεις, οι δεξιότητες, οι ικανότητες που πρέπει να διδάσκει το σχολείο. Αυτό λοιπόν ε, το διδακτικό υλικό, πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Μπορούμε να διδάξουμε το κριτικό πνεύμα, την ελεύθερη αξιολόγηση και εκτίμηση των καταστάσεων στα παιδιά και την ευθυκρισία. Νομίζω ότι αυτά που ακούσαμε μας έδωσαν μια πολύ καλή ιδέα παρά το περιορισμένο του χρόνου. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλες και όλους και τώρα θα ήθελα να δώσω νέο νέου το λόγο στους ε, δύο μιλητές. Ε, έχω όμως να πω δύο πράγματα. Πρώτον ότι η φιλανδική περίπτωση σίγουρα είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Η Φιλανδία επενδύει στην εκπαίδευση, στα ανέκπαιδευτικά συστήματα για τους δασκάλους και δίνει και ιδιαίτερη προσοχή στην έρευνα, στην παιδαγωγική επιστήμη τι πρέπει να αποφευχθεί, τι πρέπει να ενθαρρυνθεί και το καθεξής. Θα ήθελα να μου πείτε λοιπόν αν οι στρατηγικές αυτές μπορούν, οι δικές σας δηλαδή, να μεταφερθούν και να χρησιμοποιηθούν από άλλες χώρες και επίσης αν αληθεύει θέλετε να καταργήσετε τα γραπτά και όλα να γράφονται σε υπολογιστή. Αυτό με ε, δημιουργεί έτσι κάποιες, κάποια ερωτηματικά. Νομίζω ότι θα πήγαινε πολύ μακριά κάτι τέτοιο. Γιατί νομίζω ότι ε, η σκέψη και το γραπτό συνδέονται. Μιλήσατε επίσης για κάποιες υποδείξεις προς την Ευρώπη στη δική σας έρευνα. Τι ενδείξεις έχετε να δώσετε, τι μπορείτε να μας πείτε και για τις επενδύσεις και για τις στρατηγικές σας προτεραιότητες. Αυτό θα μας βοηθούσε και στη δική μας δουλειά, όπως επίσης χρήσιμο θα ήταν να μας πείτε τι θεωρείτε πιο επίγον και πιο σημαντικό σε ό,τι αφορά τους στόχους που πρέπει να τεθούν. Ευχαριστώ. 5 Πέντε λεπτά για την κάθε απάντηση, πολύ σύντομα και πιο σύντομα ή δυνατόν. Το μέγιστο, πέντε λεπτά. Ναι, ευχαριστώ, ήταν όμως τόσο πολλά τα ερωτήματα. Πολύ σύντομα. Για το γράψιμο. Ναι, η παραδοσιακή γραφή μάλλον δεν θα διδάσκεται τόσο πολύ στο σχολείο. Προσπαθούσα όμως να δείξω και από την ε, παρουσίασή μου ότι η κατάρτιση του δασκάλου ακόμα και η διδασκαλή σχολείο ασχολείται πολύ και με τα χειροτεχνικά, με τη δημιουργική ε, κίνηση και αυτό το βλέπουμε και από την ε, έρευνα σχετική με τις λειτουργίες του εγκεφάλου ότι η χρήση των χεριών και του ματιού έχει να κάνει και με τη μαθησιακή ανάπτυξη. Δεν καταργούμε λοιπόν ε, τη γραφή επειδή τη θεωρούμε πεπαλαιωμένη. Μπορεί κανείς να έχει ένα τηλεφωνάκι ή ένα μικρό υπολογιστή που μπαίνει στην τσέπη να μπορεί να τον παίρνει στην τσέπη του μέχρι και να βγει στο δάσος για τρέξιμο και να είναι όλο και πιο μικρό και να μπορεί να το χρησιμοποιήσει χωρίς δυσκολίες ε, σύνδεσης. Θέλουμε λοιπόν καινοτόμες και ευχαριστώ για την ερώτησή σας διδακτικές χρήσεις και τη λεγόμενη υβριδική μάθηση με βάση την ανάπτυξη σχεδίων. Αυθεντική τι σημαίνει μέσα, ε, έξω από την τάξη του σχολείου με καινοτόμες μεθόδους. Εγώ δεν έχω παραδείγματι κάνει κανένα μάθημα για να μάθω πώς πρέπει να χρησιμοποιώ το iPad. Μαθαίνει κανείς όμως. Και τώρα στην κατάρτιση διδακτικών των ε, μαθητές μου είναι ε, δάσκαλοι νεότεροι από την ε, κόρη μου που γεννήθηκαν μέσα στην ψηφιακή γενιά και Ε, βλέπουν ότι μπορεί η τεχνολογία να είναι και ε, φιλική ή εύχριστη ακόμα και για ξανθιές και μάλιστα άνω των 50. Μαθαίνουν λοιπόν εύκολα τη χρήση, εγώ τους δείχνω, τους μαθαίνω τη σοφία. Με αυτό το διάλογο μεταξύ γενεών μαθαίνουμε και εγώ από εκείνους όσο και εκείνοι από μένα. Πολλά μπορούμε να μάθουμε από τα παιδιά μας. Κάποιος άλλος ρωτούσε για καινοτόμες ε, παιδαγωγικές. Υπάρχουν, πιστεύω, πόροι σημαντικοί μπορεί κανείς να ζητήσει στις δραστηριότητες των ε, παιδιών και μπορούμε να μάθουμε και από τα παιδιά εάν τους δώσουμε μηχανήματα και διδαχθούμε από αυτά στη συνεργασία με άλλους μαθητές. Πολλά λοιπόν μπορούν να γίνουν ως προς την κατάρτιση των ε, δασκάλων. Βέβαια, ο κόσμος είναι γεμάτος από λάθη ή από προβλήματα που δεν μπόρεσαν να αντιμετωπιστούν. Συν το χρόνο, τα συστήματα όμως νομίζω ότι βρίσκουν αυτομάτως τη διόρθωση. Όπως γίνεται και με την επιστήμη. Κάποια στιγμή αν υπάρξει ένα λάθος στην πληροφορία που κυκλοφορεί, τα κοινωνικά δίκτυα τη διορθώνουν. Αυτή η τεχνητή ε, ευφία έχει έναν τρόπο αυτοδιόρθωσης. Και το ερώτημα εν τέλει είναι τι συμβαίνει στον κόσμο, στον πραγματικό κόσμο, γιατί για τα παιδιά αυτά, αυτός ο κόσμος είναι πραγματικός κόσμος, αυτός ο απρόσκοπτα συνδεδεμένος ευρυδικός κόσμος, συνεχίζει η ομιλήτρια και η πρόεδρος έχει ανοίξει το μικρόφωνο της. Ευχαριστώ θερμά, ο κύριος Τσό. Ευχαριστώ πολύ. Άκουσα σε αρκετά θέματα παρατηρήσεις και ερωτήσεις. Πέντε θέματα θα παρουσιάσω. Τώρα έχει να κάνει με τις επενδύσεις. Σε τι θα επένδυα. Εγώ θα επένδυα στο ανθρώπινο δυναμικό, στο προσωπικό υποστήριξης. Θα μπορεί να κάνει ό,τι μπορεί, ό,τι έχει στα, σαν δύναμη, σαν δυνατότητα ο δάσκαλος, αλλά το ίδιο και διευθυντή στις δυνατότητες που έχει στη θέση του. Γιατί μπορεί και να διδάξει, αλλά μπορεί και να παρέμβει την ώρα που είναι έτοιμο το παιδί να σηκώσει το χέρι και να χτυπήσει ένα άλλο μαθητή. Και αυτό πρέπει να γίνεται. Πρέπει να είναι παρόν αν καταραίουν τα πάντα και είναι ε, έτοιμος να διορθώσει, να συνδυάσει πληροφορία, γνώση τεχνολογίας και το καθεξής. Προσβασιμότητα, γενικά αυτό θα είναι η ηγεσία και η καθοδήγηση του σχολείου. Ε, θεματολογικά ένα άλλο κομμάτι ήταν αυτό με τις ανεπιθύμητες εκβάσεις της τεχνολογίας και την απώλεια συναισθηματικών δεξιοτήτων. Μία τουλάχιστον μελέτη που έχω υπόψη μου λέει ότι ένα παιδί που ε, στερείται ε, του μηχανήματος με το οποίο παίζει και μπει σε, σε μια κατασκήνωση μπορεί να μην έχει το ίδιο καλέ συναισθηματικέ δεξιότητες ή ότι μπορεί με το χαρτί και το μολύβι να αναπτύσσει καλύτερε. Εν πάση περιπτώσει αυτά όλα υπάρχουν πάντοτε αναστούμε καλύτερου τρόπου να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία. Τρίτο θέμα, τρίτη θεματολογική ενότητα. Τι είδου γνώση θέλουμε στη διαλειτουργικότητα τη γνώση και μάλιστα η μία διαφάνεια μιλούσε για ηθαγένεια, για πολίτη, για καλύτερη παρουσία του πολίτη στα κοινά. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μέσα και project που μπορούν να αναπτυχθούν με το iPad, με τον υπολογιστή, στοχευμένα. Φερρυπίν να ενημερωθεί ένας μαθητής, μια ομάδα μαθητών για τα προβλήματα των αστέγων ή για τη ρήπανση ή τα προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν σε κοινωνικό επίπεδο για τη φτώχεια. Όλα αυτά υπάρχουν και είναι προβλήματα της πραγματικής ζωής υπαρκτά και σημερινά και δεν χρειάζεται να περιμένουμε να βγει από το σχολείο μαθητής για να ενημερωθεί για αυτά, ούτε να πιάσει δουλειά. Θεματολογική ενότητα υπαριθμών 4. Τα λάθη που διαπιστώνονται στην πληροφόρηση μέσω του διαδικτύου. Αυτό που αναέφερε η συνάδελφος ήδη για την δικτυωμένη ευφυΐα είναι αληθές. Επίσης υπάρχει και μια ψηφιακή αλήθεια διαφορετική. Για τις ορισμένες ε, κουλτούρες ή νοοτροπίες είναι αποδεκτή η όλες όχι. Πιέζοντας όμως περαιτέρω αυτή τη λογική, βλέπουμε ότι η γνώση πιεστος ομως περαιτερω αυτη τη λογικη πολιτιστικό και κοινωνικό αγαθό περισσότερο. Παλιότερα λέγανε ότι ο άνδρας και δίλευ, της λευκής φυλής είχε το προνόμιο της, γλώσσης, της γνώσης. Τώρα είναι ξεπερασμένο αυτό. Και εν τέλει μπορώ να πω με τη συνείδηση ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της γνώσης στο διαδίκτυο είναι δικτυωμένη ευφυΐα και δεν χρειάζεται να ανησυχούμε τόσο πολύ. Τελευταία θεματολογική ενότητα. Ποιος θα διδάξει τα παιδιά τη χρήση τεχνολογία αν είναι σε θέση μόνο τους τα παιδιά. Θα έλεγα και ναι και όχι και από προσωπική εμπειρία μάλιστα. Γιατί εγώ συνεργάζομαι με φοιτητέ κάπου στα 19 και κοιτάω να δω τι είδους ε, ε, δεξιότητες μπορεί να έχουν σε γραμματιακή δουλειά που δεν τις έχουν όλες. Χρειάζεται να μάθουν, χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν ένα κείμενο ε, σε PowerPoint, να μάθουν να χρησιμοποιούν ένα κείμενο σε Word, σε PowerPoint, να ετοιμάσουν ένα πίνακα Excel. αλλά δεν τα έχουν όλα έτοιμα και πρέπει να κάνουν επιλογές. αλλά ταυτόχρονα προσπαθούμε να δείξουμε και στα παιδιά ε, γνώση που έχουν να κάνουν με την προστασία του ιδιωτικού βίου, του να μην δίνουν τι φωτογραφίε στον ε, φίλο ή τη φιλενάδα γιατί είναι προσωπικέ και μπορεί αυτό μετά να πάει να τι πουλήσει στο δίκτυο και το καθεξή. Αυτά που έχουν να κάνουν με την κοινωνική ευφία. Σα ευχαριστώ πολύ. Έχουμε καθυστερήσει. Θα δώσω το λόγο τώρα, ζητώντας παρακαλώ να είσαστε σύντομοι και να λάβετε υπόψη σας και τις ερωτήσεις τις οποίες ε, σας δείξαμε. Οι χρήστες ε, ψηφιακών υπηρεσιών από δορυφορική πηγή. Δέκα λεπτά παρακαλώ, γιατί αλλιώς φοβάμαι ότι θα ε, μείνουμε πίσω. Okay. Um, thank you very much, Madam Costa, for inviting me the committee today. It's uh, my privilege to be here. Um, Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε να μιλήσω εδώ. Εκπροσωπώ την ΕΣΟΑ, μια ένωση που εκπροσωπεί ε, τους ε, δορυφορικούς ε, παρόχους υπηρεσιών και άλλες εταιρείες βέβαια που παρέχουν ε, υπηρεσίες επικοινωνίας και στα κράτη-μέλη της Ένωσης, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Φαντάζομαι ότι πολλοί από εσάς στην αίθουσα διερωτάστε ε, γιατί σε αυτή τη συζήτηση για τη διεθνή στο σχολείο μιλάμε για τους δορυφόρους. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω με λίγα λόγια ως προς αυτό το σημαντικό με τους ε, είναι ότι μπορούν να φτάσουν και να διασυνδέσουν τον κόσμο εξάτω του που μένει. Αν μένουν σε νησιά, σε βουνά, σε κοιλάδε, σε παιδιάδε, σε πολύ ε, απομονωμένες ε, ε, υβαλτόδε περιοχέ κτλ. Παρόλα αυτά μπορούν να συνδεθούν όλοι με το δορυφόρο και η διασύνδεση αυτή να γίνεται ζήτημα ημερών. Χρειάζεται απλά ένα πιάτο και ένα μόντεμ αν το πιάτο ε, το εγκαταστήσετε σε οποιοδήποτε κατάστημα, βιβλιοθήκη, νοσοκομείο, σχολείο, ε, ακόμη και στη μέση, στην πλατεία μιας ε, μικρής κοινότητας ενός χωριού που μπορεί να ε, έχει ε, να σου δώσει μέσα σε λίγε ημέρε ε, μία λύση υψηλή τεχνολογία Από οικονομική πλευρά είναι προσιτό. Ναι, είναι και θα σα δώσω ένα παράδειγμα από την Ιταλία. Για εσά, κυρία Κώστα, αφιερωμένο. Εδώ βλέπετε από ένα από τα μέλη μα, 22 Mbit το δευτερόλεπτο είναι η προσφορά, με μηνιαία συνδρομή και για 25 ευρώ το μήνα συγκεκριμένα. Πρόκειται για μια προσφορά διασύνδεσης ε, στο διαδίκτυο για τι αγροτικέ περιοχέ ή τι πραστιακέ περιοχέ, κάτι το οποίο διατίθεται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Άρα, πραγματικά πολύ λίγοι είναι οι λόγοι ή οι δικαιολογίε να πει κανείς ότι εξακολουθεί να δικαιολογείται πράξη ένας ψηφιακού χάσματο στην Ευρώπη. Η Κομισιόν να γνωρίζει ε, ήδη από το 2013 την σημασία τη, των δορυφόρων και μας ζήτησε να συνεισφέρουμε, να έχουμε μέχρι το 2013 100% ευρυζωνικής ε, διασύνδεσης. Με ε, τον κύριο Βιόλα από την Γαμαλίτα Connect ε, θελήσαμε να αναπτύξουμε ένα εργαλείο το οποίο ξεκίνησε εδώ το Νοέμβριο του 2013 με τον κύριο Φανίλη Στερό και λέγεται Broadband for All. Εάν κλικάρετε πάνω σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ένωσης θα βρείτε στη γλώσσα της χώρας ε, τον κατάλογο των διανομέων των αντιπροσώπων που μπορούν να διασυνθέουν τους χρήστες όπου και αν αυτοί βρίσκονται. Μιλάμε λοιπόν τώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε πράγματι 100% ευρυζωνική κάλυψη, ε, αγωνιστήκαμε από κοινού, έχουμε τα εργαλεία στη διάθεσή μα. Όταν μιλάμε για την ίδια την σύνδεση, ε, εκεί έχουμε πρόβλημα. Το 63% των 9χρονων δεν έχουν ψηφιακό εξοπλισμό και πρόσβαση σε αυτόν στα σχολεία. Ξέρουμε ότι 50 με 80% των μαθητών δεν έχουν ποτέ χρησιμοποιήσει ε, textbook ή παιχνίδια εκπαιδευτικά ή διάφορα λογισμικά ε, για να λύνουν ασκήσεις σε ηλεκτρονική μορφή. Παρ' όλα αυτά λοιπόν και παρά τις δεσμεύσεις ε, δεν ε, έχουμε παρά ένα πολύ μεγάλο ακόμη ψηφιακό χάσμα ψηφιακή, μάλλον δορυφορική ευρυζωνικότητα δεν είναι κάτι καινούργιο. Ίσως το ακούτε εδώ ε, ορισμένοι για πρώτη φορά, αλλά υπάρχει εδώ και κάποια χρόνια και έχουμε εκατοντάδε. χιλιάδες διασυνδεδεμένου χρήστες στην Ευρώπη. Έχουμε όμω και δορυφορικέ λύσεις για τα σχολεία. Θα ήθελα να σας δώσω δύο σύντομα παραδείγματα από τη Γαλλία και τα δύο γιατί με την εμπειρία μας βλέπουμε ότι η Γαλλία ως κράτος μέλος έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία στη χρήση ανάπτυξη της δορυφορικής ευρυζωνικότητας και βλέπετε πώς μπορεί κανείς να είναι δημιουργικός. Αυτό είναι από μια ε, θεωρία που λέγεται VVOL, ecolconnecte.fr και εδώ βλέπετε ένα παράδειγμα του πόσο κοστίζει. Και μετά η εταιρεία Nordnet, Connect Call, αυτό το παράδειγμα έχει το καλό ότι στα δεξιά βλέπετε ένα μικρό τετραγωνίδιο ακριβώς από πάνω, ε, από την διασύνδεση που σου λέει πώς μπορείς να ε, βοηθηθείς. Λέει η Net Financière proposée par l'État. Το κράτο προτείνει χρηματοοικονομική βοήθεια, επιδοτήσει, χωρί τα λοιπά. Πολλοί δεν έχουν πληροφορίε, δεν ξέρουν ότι υπάρχει λύση, αλλά δεν ξέρουν ότι μπορεί και να του δοθεί δωρεάν η υπηρεσία, δηλαδή να επιστραφεί το κόστο. Βλέπουμε λοιπόν πλέον ότι ζούμε ε, σε μια εποχή που μπορεί να υπάρξει κατανόηση περιεχομένου σε οποιαδήποτε συσκευή, τεράστιο δυναμικό βελτίωση ε, τη εκπαίδευση που λαμβάνουν ε, οι Ευρωπαίοι μαθητέ, προσφέρει αυτή η τεχνολογία. Αλλά πρέπει να δούμε ότι τα παιδιά μας ήδη από σήμερα έρευνουν στο ίντερνετ, ανεβάζουν τις εργασίες τους στον υπολογιστή, κάνουν τα project συνεργαζόμενοι μέσω υπολογιστών, βλέπουν ηλεκτρονικά βιβλία, βίντεο και μάλιστα site όπως το mathletics.com ε, μπαίνουν τα παιδιά από διάφορες χώρες του κόσμου σε αυτά τα site ε, και ε, λύνουν ασκήσεις κτλ. Πρέπει να προσπαθήσουμε όλη αυτή την πρόσβαση σε αυτά τα δίκτυα να την καταστήσουμε δυνατή για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και περιφέρειες. Και εδώ οι δορυφόροι είναι κλειδί γιατί μπορούν να βοηθήσουν ε, αυτούς που δεν, ε, τα σχολεία που δεν έχουν οπτικές σύνες, DSL κτλ. Ξέρουμε παραδείγματος χάρη στην Γαλλία ότι 17.000 σχολεία δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Γνωρίζουμε επίσης ε, ότι μια εικόνα αξίζει ως χίλιες λέξεις. Και ξέρουμε ότι τα σχολεία όλο και περισσότερο χρησιμοποιούν πιο εξειδικευμένα βοηθήματα για την διδασκαλία. Αυτό το περιεχόμενο νομίζω ότι είναι ιδανικό για να μεταδοθεί μέσω δορυφόρου. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο σημαντικό κομμάτι στην εξίσωση αυτή. Είναι η διδακτέα ύλη των σχολείων πολύ σημαντική πληροφορία, την ξέρουμε εκ των προτέρων και αν δώσουμε και στους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου αυτές τις πληροφορίες μπορούν αυτοί να αναπτύξουν προϊόντα προσαρμοσμένα, εξατομικευμένα ανάλογα με τη δακτέλη του κράτους μέλους ή το κράτος μέλος. Αν έχουμε λοιπόν αυτή τη δυνατότητα διασύνδεση με την τεχνολογία τη δορυφορική μπορεί να κάνει ε, κανείς πιο ε, αποδοτικά, αποδοτική τη διαδικτύωση και θα μπορούν να μεταφορτώνουν τα παιδιά πολλά εργαλεία για να μπορούν να ζήσουν μια πολύ πιο ταχεία και οικοδομητική διδακτική εμπειρία. Ολοκληρώνοντα, σας ρωτώ, έχετε γνωρίσει ποτέ ένα παιδί που να μην το συναρπάζει το διάστημα, να μην το συναρπάζει το ότι ε, ε, έχουμε προσελεινωθεί, ότι και πρόσφατα προσγειωθήκαν πάνω στη, σε ένα κομίτι και το καθεξής. Ε, έχουμε ε, τη δυνατότητα των δορυφόρους να αγγίξουμε, να έχουμε πρόσβαση στη ζωή εκατομμυρίων. Ε, ξέρω ότι όλοι παρακολουθείτε ότι γίνεται στο Νεπάλ η προσπάθεια ανοικοδόμησης, ανακούφισης, αλλά αυτό μπορεί να γίνει το δίκτυο, όπως μπορεί να γίνει και η απλή επικοινωνία με το Skype, Άρα ο δορυφόρος πραγματικά μπορεί να αγγίξει τις ζωές όλων και να φτάσει σε σημεία που μπορεί να φτάσει εύκολα άλλη τεχνολογία. Η ΕΣΟΑ είμαστε στη διάθεσή σας να συνεργαστούμε με την Κομισιόν και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε όλες οι βάδιθες σας να γίνουν ψηφιακές. Thank you so much. Very interesting, very... Σας ευχαριστώ για μια πολύ ενδιαφέρουσα και συγκινητική παρουσίαση θα έλεγα. για τον ρόλο τον οποίο ήδη παίζει ο δορυφόρος για τη σύνδεση των σχολείων στην Ευρώπη. Θα δώσω τώρα το λόγο τον Όμπετ Τιούμπνα, υπεύθυνο της ΙΖΑ για τα καινοτόμα σχολεία από πλευράς της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. εκπροσωπώ τις τηλεπικοινωνίες της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας και του Τμήματος Εφαρμογών. Θα ξεκινήσω με κάποιες εισαγωγικές παρατηρήσεις. Να σας πω ότι εμείς δεν ασχολούμεθα μόνο με τις τεχνολογίες αλλά και τις εφαρμογές. Έχουμε 22 χώρες μέλη, η Ουγγαρία και η Εστονία μόλις έγιναν μέλη και ο Καναδάς συμμετέχει στα πλαίσια μια συμφωνίας συνεργασίας. Η πλειοψηφία των προγραμμάτων μας είναι εθελοντικά προγράμματα. Οι χώρες ανάλογα με την επιθυμία τους συμμετέχουν εκτός από την εξερεύνηση του αποτάτου διαστήματος και του ηλιακού συστήματος, εκεί η συμμετοχή όλων των χωρών είναι υποχρεωτική. Εδώ είναι οι προπολογισμοί μας, Βλέπετε ότι συνολικά μιλάμε για 4 δις 400 εκατομμύρια. Ε, για τις εφαρμογές ξοδεύουμε κάτω των 40 εκατομμυρίων κατέτος και τα υπόλοιπα πηγαίνουν στην ανάπτυξη των τεχνολογιών υποδομής για το διάστημα. Τώρα σε πιο συγκεκριμένες εφαρμογές. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι προγράμματα υποδομών τα πράσινα που βλέπετε είναι εφαρμογές επικοινωνίας ε, με δορυφόρους, μέσω δορυφόρων και ενσωματωμένες ε, εφαρμογές και προώθηση αυτών των ε, ενσωματωμένων εφαρμογών όπως οι γεωδεσικοί παρατηρητές και η παρατήρηση του διαστήματος. Έχουμε αλλάξει τις δραστηριότητες σε σχέση με το παρελθόν. Βλέπουμε εδώ ποιος είναι ο στόχος μας, ποιοι είναι οι χρήστες, η κοινότητα η οποία απαιτεί κάποιες, έχει ανάγκη κάποιες υπηρεσίες. Και για να γίνει αυτό απαιτούνται κάποιες ε, τεχνολογίες. Πρόκειται για ένα πολυεπίπεδο θα έλεγα έτοιμα αν θέλετε από πλευρά ε, των κοινοτήτων, θέματα εκπαίδευσης, Βέβαια οι δραστηριότητες μας είναι πολύ μικρές στον τομέα της εκπαίδευσης σε σχέση με τις άλλες δραστηριότητες. Βλέποντας τα θέματα τώρα της συνδεσιμότητας στην Ευρώπη με το ευρύ φάσμα, βλέπετε ποιος είναι ο στόχος για το 2020. Η μεγάλη πλειοψηφία των χωρών δεν θα είναι απόλυτα συνδεδεμένες. Κάποιες χώρες ακόμα δεν έχουν διευκρινίσει τα επίπεδα συνδεσιμότητας τα οποία επιθυμούν. Συλλέγουμε πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Απαιτούνται περαιτέρω επενδύσεις, ισχυρές επενδύσεις, οι οποίες αφορούν κυρίως επίγειες υποδομές, όπως είναι ψηφιακές κτλ οι δορυφορικές υπηρεσίες βοηθούν με εύκολο τρόπο τις επικοινωνίες. Ξέρετε το παράδειγμα της Αυστραλίας που είναι έτοιμη να συνδέσει τους δορυφόρους παρατήρησης που έχει με τα δίκτυα τηλεπικοινωνίας. Στο παρελθόν προωθήσαμε αρκετά προγράμματα με αρκετή επιτυχία ανάλογα. Θα σας αναφέρω ορισμένα από αυτά. και μπορείτε να πάρετε τις παραπομπές ακριβώς για το πώς το έχουμε πετύχει. Βλέπουμε τις επιπτώσεις της των εφαρμογών αυτών, όχι μόνο σε τεχνολογικό επίπεδο. Εμείς παρέχουμε την τεχνολογία, το περιεχόμενο και ταυτόχρονα ε, προχωράμε σε πιλωτικές ενέργειες, σε πιλωτικές δράσεις. Δύο παραδείγματα. Καταρχάς, ε, μια εφαρμογή για τα παιδιά, για τα σχολεία μάλλον, μέσω των τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι υπηρεσίες εξακολουθούν να παρέχονται, αλλά με το πέρασμα των χρόνων οι τεχνολογίες SATCOM έχουν αντικατασταθεί από επίγεια δίκτυα με, με ίνες και έτσι εμείς ήμασταν το κύριο μέσο αν θέλετε, αλλά τώρα έχουμε αντικατασταθεί. Ένα πρόσφατο είναι η εξαποστάσεως ε, ε, μαθητεία. Εδώ παίζει μεγάλο ρόλο ο ανθρώπινος παράγοντας φυσικά. Μπορούν οι γιατροί σαν παράδειγμα να μάθουν πάρα πολλά από ε, ομολόγους τους, αλλά δυστυχώς το σχέδιο δεν προχώρησε, απέτυχε θα έλεγε κανείς οι γιατροί προτιμούσαν να πηγαίνουν σε συνέδρια ή να κάνουν πρακτική μαθητεία σε διαφορετικά επίπεδα. Έχω επίσης και κάποια άλλα παραδείγματα του πρόσφατου παρελθόντος της χρήσης των δορυφόρων για την εκπαίδευση στην Νότια Αφρική σαν παράδειγμα. Το θέμα ήταν να δείξουμε στους ε, καθηγητές και δασκάλους πως να μάθουν να μεταδίδουν τις ε, γνώσεις τους και τις ικανότητές τους μέσω του διαδικτύου φυσικά και των ε, δορυφορικών δικτύων. Και όχι μόνο μέσα στο σχολείο, αλλά και στα κοινοτικά καφέ εκτός σχολείου. Ε, υπάρχουν επίσης και νέες πλατφόρμες εκμάθησης και ενωτόμες αυτή τη φορά, με ε, μέσα και οι ίδιοι οι καθηγητές και οι μαθητές είναι και δημιουργοί του περιεχομένου της διδακτικής ύλη. Βλέπετε κάποιες φωτογραφίες που έχουν σχέση και με τις προηγούμενες ομιλίες οι εφαρμογές αυτές των ψηφιακών τεχνολογιών δεν είναι κάτι το πάρα πολύ εύκολο. Ε, χρειάζονταν 400 δολάρια σαν παράδειγμα το μήνα για τα σχολεία για να μπορούν να λειτουργούν με τον τρόπο αυτό. Αλλά παρόλα αυτά διευκολύναμε ε, πολύ την ε, διεύρυνση των δικτύων αυτών των μαθησιακών στην Αφρική δεν είναι ένα πράγμα σπάνιο και μαγικό. Υπάρχει, αρκεί κανείς να οργανώσει έναν διαγωνισμό και θα υπάρξουν προσφορές από διάφορους παροχής υπηρεσιών, ψηφιακών διαστημικών υπηρεσιών, δορυφορικών συγγνώμη υπηρεσιών. Συμπερασματικά τώρα, Νομίζω ότι τα SATCOM, οι δορυφορικές επικοινωνίες, μπορούν πολλά να προσφέρουν στην εκπαίδευση. Βέβαια οι επίγειες ε, μέθοδοι επικοινωνίας είναι ευθυνότερες και πιο πρακτικές. Αυτό το οποίο απαιτείται στον τομέα της εκπαίδευσης είναι η παροχή υπηρεσιών SATCOM. Αυτό είναι το εύκολο κομμάτι, υπάρχει τεχνολογία. Το πιο δύσκολο είναι να δημιουργηθεί πραγματικό περιεχόμενο και το περιεχόμενο αυτό να διανεμηθεί σωστά και να είναι πιστικό και εύχριστο. Έτσι θα διευκολύνουμε την απορρόφηση των νέων αυτών τεχνολογιών στις απότερες απομεμακρυσμένες περιοχές. Και εδώ τίθεται το θέμα του ανθρώπινου παράγοντα. Σας έχω πει ότι τεχνολογίες υπάρχουν εδώ και 5-6 χρόνια. Απαιτείται όμως ε, κάτι παραπάνω, υπάρχει το θέμα του κόστους, και η προσφορά που υπάρχει είναι δεδομένη, έχετε εδώ κάποια παραδείγματα. Για το εκπαιδευτικό περιεχόμενο είδαμε εμείς στα προγράμματά μας ότι υπάρχει μία μετακίνηση από το γραμμικό σύστημα διδασκαλίας σε ένα σύστημα όπου η δημιουργία περιεχομένου με πολυμέσα γίνεται και από τους καθηγητές και από τους μαθητές η χρήση και η αποδοχή των συστημάτων αυτών εξαρτάται από τον ανθρώπινο παράγοντα και από τον τεχνολογικό παράγοντα. Για να συναντηθούν με σωστό τρόπο οι δύο αυτοί παράγοντες απαιτείται ε, προσπάθεια και προσοχή για μια καλή επικοινωνία και οι πολίτες, ε, ο ανθρώπινος παράγων να νιώθει ότι ελέγχει το σύστημα, ότι είναι εξοικειωμένος και του ανήκει το σύστημα. Αυτά τα οποία έχουμε κάνει σε διάφορες περιοχές σε μικρή κλίμακα είναι κάτι το οποίο μπορεί να διευρυνθεί όχι μόνο οι διδάσκοντες αλλά τεχνική υποστήριξη, οργάνωση και στο τέλος το θέμα των δωρητών και αυτών που καλύπτουν το κόστος. Τώρα για τις μελλοντικές χρήσεις βλέπετε εδώ οι δυνατότητες αύξησης της χρήσης του διαδικτύου στο μέλλον Υπάρχουν ε, διάφορες προτάσεις, ο Μπράνσον και άλλοι θέλουν να θέσουν σε κυκλοφορία χαμηλού ύψους χιλιάδες δορυφόρους έτσι ώστε να παρέχουν δορυφορικές συνδέσεις διαδικτυακού τύπου σε όλο τον κόσμο. Αυτό ε, είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά μελλοντολογικό. Δεν ξέρω τι εξελίξεις ε, χρειάζονται σε τεχνολογικό επίπεδο και επίσης και τι θα γίνει τελικά και πώς θα χρησιμοποιηθεί η συνδεσιμότητα η οποία θα είναι διαθέσιμη. Τεράστιες ταχύτητες κυκλοφορίας δεδομένων, δεκαπλάσιες των διαθεσίμων σημερινών ανωτάτων ταχυτήτων. Απίστευτα πράγματα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ, λέει η κυρία Κώστα. Ήδη εσείς έχετε ανοίξει εδώ κάποιες δυνατότητες πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Περνάμε τώρα στον Τζοβάνι Μπιόντι. Θα πω ότι εδώ και δέκα χρόνια η Ινδία ξεκίνησε με έναν δορυφόρο εκπαιδευτικό για να ξεπεράσει τα κενά τα οποία υπήρχαν σε επίπεδο εκπαίδευσης στην Ήπεθρο, κάτι το οποίο βοήθησε να καλυφθούν πολλά από τα κενά αυτά. Περνάμε τώρα στον καθηγητή Τζοβάνι Μπιόντι, πρόεδρο του Schoolnet, του Ευρωπαϊκού Δικτύου Σχολείων, ή Σχολικού Δικτύου. Ευχαριστώ, καλημέρα σας. θα εκπροσωπήσω το δίκτυο των σχολείων και να δώσω ίσως και κάποιες απαντήσεις στα ερωτηματικά που τέθηκαν. Το δίκτυο δημιουργήθηκε εδώ και 20 περίπου χρόνια μετά από μια πρωτοβουλία των Υπουργών Παιδείας. Στην παρούσα φάση συγκεντρώνει την συνεργασία 30 Υπουργείων. Όλα τα σχέδια του Ευρωπαϊκού Δικτύου Σχολείων επηρεάζουν άμεσα θα έλεγα όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς. Αυτό το αποδεικνύουν οι αριθμοί αν θέλετε. Έχουμε το twinning με 310.000 εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν. Έχουμε επίσης και θεματικά επίπεδα όπως η ασφάλεια των δικτύων, οι θετικές επιστήμες. Ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα επίσης αναδιοργάνωση ε, των μελλοντικών σχολικών τάξεων. Τι μπορεί να είναι το μέλλον ενός σχολείου, πώς μπορεί να αλλάξει το σχολείο μέσω των τεχνολογιών και μέσω μιας πραγματικής υποστήριξης για καλύτερη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Εδώ και δεκαετίες είχε δημιουργηθεί μια δικοματική επιτροπή στο Κογκρέσο για να δούμε αν μπορεί να αλλάξει το διαδίκτυο τα σχολεία. Και η απάντηση ήταν καταφατική. Το θέμα είναι αν τα σχολεία είναι σε θέση να περάσουν σε αυτές τις αλλαγές, αν έχουν καθυστερήσει τα σχολεία αυτή τη διαδικασία, αν έχουν υπάρξει αντιστάσεις για την δυνατότητα αυτή. Να πω επίσης ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης που προηγήθηκε μιλήσαμε για τεχνολογίες, θεωρώντας ότι οι τεχνολογίες αυτές είναι βασικά το ίντερνετ. Θα ήθελα όμως να θυμίσω σε όλους ότι το σχολείο είναι γεμάτο από τεχνολογίες. Η γραφή είναι τεχνολογία, το βιβλίο, το στυλό, το μολύβι. Και όλες αυτές είναι τεχνολογίες με τις οποίες έχουμε συνηθίσει, δεν τις θεωρούμε κάτι το περίπλοκο, είναι τμήμα της καθημερινότητάς μας. Γιατί εμείς που ερχόμαστε από μία γιανιά ε, που ονομάζεται τώρα πλέον οι ψηφιακοί μετανάστες ε, για τα παιδιά μας, να μην ξεχνάμε, το υπολογιστής είναι ένας φίλος απλά, όπως ήταν για μας το βιβλίο. Λοιπόν, προχωράω με το δίκτυο. Το κεντρικό θέμα το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας είναι η αλλαγή του σχολικού προτύπου. Δεν υπάρχει ψηφιακό σχολείο. Υπάρχει το σχολείο. Το σχολείο μπορεί να χρησιμοποιήσει τις τεχνολογίες για να μετασχηματίσει ένα μοντέλο, ένα πρότυπο. Τον προηγούμενο αιώνα Τα μεγάλα συστήματα τα εκπαιδευτικά είχαν σαν κεντρικό θέμα το θέμα του αλφαβητισμού του μεγάλου τμήματος του πληθυσμού που συνδεόταν με τη βιομηχανική επανάσταση. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, έχουν αλλάξει οι στόχοι γιατί τώρα έχει αλλάξει η κοινωνία. Είμαστε μια κοινωνία γνώσης και περνάμε από τη διδασκαλία στην εκμάθηση. Δεν είναι δευτερεύον αυτό. Πρέπει να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο εκμάθησης, πρέπει να αλλάξουμε το σενάριο λειτουργίας του σχολείου. Τα παιδιά πρέπει να γίνουν πρωταγωνιστές στην οικοδόμηση της δικής τους γνώσης. Και αυτό σήμερα είναι δυνατό, αυτό σήμερα είναι εφικτό, λόγω και χάρη στην ψηφιακή γλώσσα. Μιλάμε για το διαδίκτυο, σκεφτείτε το Wikipedia, σκεφτείτε το ότι τα παιδιά μας ε, συλλέγουν τεράστιες πληροφορίες. Ο ψηφιακός χώρος σήμερα ε, δίνει την δυνατότητα εργαστηρίων ψηφιακών, δίνει τη δυνατότητα της εξομοίωσης και του ελέγχου σε πραγματικό χρόνο των ερευνών και των διαδικασιών. Περνάμε από τον ε, καθηγητή που περιγράφει έναν πυρήνα με τη μετακίνησή μας μέσα σε έναν πυρήνα. Ε, κάποιον ο οποίος περιγράφει το ηλιακό σύστημα σε κάποιον ο οποίος μπαίνει μέσα στο ηλιακό σύστημα. Αυτές είναι οι δυνατότητες που δίνει ο ψηφιακός κόσμος στο σχολείο. Προσπαθούμε να καταστήσουμε τη διαδικασία της εκμάθησης διαλειτουργική. Τα παιδιά γίνονται πρωταγωνιστές της διαδικασίας της μαθησιακής βιώνουν με ευτυχία το χρόνο τους στο σχολείο, είναι πρωταγωνιστές. Όταν τα παιδιά βγαίνουν από το δωμάτιό τους στο σχολείο, είναι πρωταγωνιστές του ψηφιακού τους κόσμου, οικοδομούν τον κόσμο των γνώσεών τους, οικοδομούν αν θέλετε τον δικό τους μουσικό κόσμο Αυτό το οποίο κάνουμε εμείς λοιπόν σαν Ευρωπαϊκό Δίκτυο είναι να υποστηρίξουμε και να παρέχουμε ένα πλαίσιο σε αυτές τις αλλαγές. Αυτό το κάνουμε και βοηθώντας τους εκπαιδευτικούς, βοηθώντας την κατάρτισή τους, βοηθώντας επίσης την συνεργασία αυτών οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο πρέπει να λειτουργήσουν ηγετικά, συντονιστικά σε σχολικό επίπεδο ενισχύουμε τη δημιουργία δικτύων ανάμεσα σε σχολεία, ενισχύουμε τη συμμετοχή τους στα ευρωπαϊκά ταμεία και μέσα που είναι ένα σημαντικός τρόπος για μας έτσι ώστε να πετύχουμε κάποιες από τις πρωτοβουλίες τις οποίες θέλουμε να προωθήσουμε. Μία από τις πρωτοβουλίες αυτές είναι η δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ακαδημίας, μιας Ακαδημίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι αλήθεια ότι για να επενδύσει κανείς σε τεχνολογίες πρέπει να επενδύσει σε ανθρώπινο δυναμικό. Και αυτό είναι ουσιώδες. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκού επίπεδου ακαδημία η οποία με εγκάρσιο τρόπο θα στηρίξει όλες τις διαδικασίες αλλαγής του μοντέλου, δηλαδή μελλοντικέ τάξεις, αναδιοργάνωση χωρική. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία, στα οποία μπορούμε να βοηθήσουμε. Εμείς μέσω της δικτύωσής μας παρέχουμε ένα πλαίσιο συνεχούς κατάρτισης των διδασκόντων. Αναφέρομαι εδώ στην Ιταλική κατάσταση στην παρούσα φάση. Ιδιαίτερα στα πλαίσια της διαγενεϊκής διαδοχής των διδασκόντων βελτιώνεται η γνώση του ψηφιακού κόσμου και διαμορφώνεται μια καλύτερη εικόνα των αλλαγών που θα βιώσει και που βιώνει το σχολείο. Εδώ να πω και κάποιους αριθμούς. Εμείς κάναμε και κάποιες εμπειρίες δημιουργώντας κάποιους πυρήνες με 3.000 εκπαιδευτικούς σαν παράδειγμα οι οποίοι πήραν την πρωτοβουλία να εγγραφούν σε μικρά προγράμματα, 1.600 σχολεία, είναι μικροί αλλά σημαντικοί αριθμοί που δείχνουν ότι υπάρχουν ανάγκες από πλευρά των σχολείων. Αυτά τα κάναμε δυστυχώς μόνο στα αγγλικά για λόγους ανάγκες. Θα θέλαμε ε, τα μαθήματα αυτά να γίνουν και σε άλλες γλώσσες, γιατί η μοναδική χρήση της αγγλικής είναι πολλές φορές ένα εμπόδιο για τους καθηγητές. Ένα άλλο θέμα στο οποίο θέλουμε να επενδύσουμε είναι η δημιουργία μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης. Εκεί μπορούμε να ανταλλάξουμε το περιεχόμενο που παράγουν οι ίδιοι οι διδάσκοντες. Η πραγματική διδακτική ύλη δηλαδή η οποία οφείλεται στις διαφορές των εκπαιδευτικών μας συστημάτων που οδηγεί σε διαφορετικά περιεχόμενα. Ε, και για την, ε, τον τομέα των κυτάρων, των πυρήνων, τον τομέα των εξισώσεων δευτέρου επίπεδου. Βλέπουμε ότι οι εκπαιδευτικοί παράγουν περιεχόμενο, παράγουν ε, πράγματι ενδιαφέροντα, ενδιαφέρουσες προτάσεις και δημιουργούν μια κληρονομιά η οποία θα πρέπει να ενταχθεί σε ένα ενιαίο σύστημα. Η τελευταία παρέμβαση αφορά την δορυφορική δικτύωση. Το θέμα είναι με αυτό να στηρίξουμε τα μικρά σχολεία. Σχολεία τα οποία μόνο λόγω της ε, τεχνολογίας θα παραμείνουν ε, διαδικτυωμένα. Ορεινές περιοχές, νησιωτικές περιοχές που θα μπορέσουν να διευρύνουν όχι μόνο το γνωσιακό τους περιεχόμενο και περιβάλλον αλλά και το κοινωνικό τους περιβάλλον. Όταν είναι, είμαστε λίγοι καταλαβαίνετε ότι οι απομακρυσμένες περιοχές δεν θα τα καταφέρουν πολύ καλά όπως δείχνουν και οι μελέτες του ΟΣΑ. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο μικρών σχολείων, δίκτυο το οποίο θα συμμερίζεται πρότυπα αηφορίας και τα οποία θα δίδουν εγγυήσει ε, για την ε, επιβιωσιμότητά τους λόγω των νέων τεχνολογιών έγιναν επιμέρους προτάσεις από πλευράς του δικτύου μας προς την κατεύθυνση αυτή σε συνεργασία με τις Γενικές Διευθύνσεις της Κομισιόν. Σας ευχαριστώ λέει η κυρία Κομπόστα. Είναι, για, είναι μια πολύ σημαντική παρέμβαση, πράγματι αφορά 30 χώρες, πάνω από 30.000 σχολεία, πλούσιες εμπειρίες και η ιδέα της Ακαδημίας και η ιδέα της βιβλιοθήκης είναι σωστές ιδέες για μας και είναι επιλογές και για τα πιλωτικά μας προγράμματα. Θα προσπαθήσουμε τις προτάσεις αυτές να τις ευνοήσουμε στο μέλλον. Θα δώσω τώρα το λόγο στους δύο γενικούς διευθυντές Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Μονέ και μετά με τον κύριο Βιόλα. Ευχαριστώ. Ναι, σχεδόν έχουμε ξεκινήσει το χρόνο μας. Τα πολλά έχουν καλυφθεί. Θα είμαι σύντομος. Εδώ δίπλα μου κάθεται ο Ρομπέρτο Βιόλο, συνάδελφος. Σύμπτωση μόνο. Μόνο και μόνο επειδή είχατε την καλοσύνη να μας προσκαλέσετε και τους δύο. Εδώ βρισκόμαστε γιατί όπως είδαμε όλο το απόγευμα δεν είναι δυνατόν να κοιτάξουμε τη σχέση μεταξύ τεχνολογίας και εκπαίδευσης χωρίς να κοιτάξουμε παράλληλα και δύο πολύ σημαντικά θέματα, την συνδεσιμότητα αλλά και παράλληλα την παιδαγωγικά σημαντική χρήση της τεχνολογίας. Στις δύο αυτές πτυχές λοιπόν μπορούμε να προσφέρουμε υπηρεσία. Ο Ρομπέρτο θα μιλήσει για τη συνδεσιμότητα, εγώ επιτρέψτε μου να περιοριστώ στην παιδαγωγική πτυχή. Ένα πράγμα που πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι η ταχύτατη ρυθμή αλλαγής πριν από δύο δεκαετίες ίσα ίσα είχε αρχίσει το Facebook. Τώρα έχει εκατομμύρια συνδεδεμένους χρήστες. Ε, ωστόσο πρέπει να δούμε την πτυχή των υποδομών, πώς μπόρεσαν αυτές να προσαρμοστούν έχετε τις αλλαγές και επίσης να δούμε πόσο δύσκολο είναι σε θέματα τόσο περίπλοκα όσο τα εκπαιδευτικά συστήματα να εισαχθούν ε, ουσιαστικές αλλαγές. Εντυπωσιακό επίση είναι το γεγονό ότι πολλοί από του ομιλητέ και μάλιστα αναφέρουμε στη φιλανδική εμπειρία ε, καταλήγουν στο συμπέρασμα όπω και η υπηρεσία μελετών του Κοινοβουλίου εν τέλει κάθε αλλαγή έχει να κάνει με ανθρώπου και το κέριο ζήτημα είναι να δοθούν στου δασκάλου τα κατάλληλα εργαλεία να μπορέσουν να αξιοποιήσουν ε, κέρια, χρήσιμα, ενδιαφέροντα εργαλεία τεχνολογίες. Πώς θα υποστηρίξουμε τους δασκάλους με το ζητούμενο. Και πριν περάσω σε αυτό, δεν θέλω να αναφερθώ σε ένα σημείο το οποίο δεν έχει καλυφθεί ακόμη, που όμως έχει κρίσιμη σημασία για μένα, εάν θέλουμε να επιφέρουμε κάποια αλλαγή στην τεχνολογία και την κερατομία. Πολύ σημαντική λοιπόν είναι η φύση της γνώσεως. Αν κοιτάξουμε τη γνώση όπως τη βλέπουμε σήμερα, γνώση δεν είναι μόνο μετάδοση πληροφορίας. Γνώση δεν είναι μόνο ε, διανομή πληροφορίας. Είναι δίκτυο, συνεργασία για το μέλλον λοιπόν σημασία έχει το συνεργατικό έργο όλο και πιο περίπλοκων δικτυωμένων ομάδων, πανεπιστημίων, κέντρων ερευνητικών κτλ. Και η διάδοση της γνώσης. Αν δούμε στα πανεπιστήμια, η δικτύωση έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί τα πανεπιστήμια δεν είναι διατομεακά, δεν είναι ευέλικτα, δεν είναι σε θέση να εργάζονται σε δύσκολα και αβέβαια περιβάλλοντα. Άρα κρίσιμη σημασία στο ευρωπαϊκό επίπεδο θα είναι να εισαχθεί ο εξυγχρονισμός των εκπαιδευτικών συστημάτων στο θεματολόγιο για την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μία έκκληση που μπορώ ταπεινά να απευθύνω στην Επιτροπή σας είναι να υπάρξει θέση για την εκπαίδευση στη μελλοντική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη δάσλος θα έχουμε χάσει το τρένο και δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Δεν θα έχει δε, ούτε και θα έπρεπε να έχει ρυθμιστικές και κανονιστικές εξουσίε στον χώρο τη εκπαίδευση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει λοιπόν την καινοτομία και την αλλαγή στα εκπαιδευτικά ιδρύματα να την προαγάγουμε. Αυτό είναι το κρίσιμο ζητούμενο έτσι ώστε η τεχνολογία όπω και στου άλλου τομεί να αποτελέσει όφελος και για την εκπαίδευση. Ε, να μιλήσω τώρα για τους εκπαιδευτές και τους ε, διδασκάλους. Αν κοιτάξουμε λοιπόν, το τι γνωρίζουμε για τους δασκάλους. Οι δάσκαλοι μας λένε δύο πράγματα. Το ένα είναι το τι χρειάζονται, ξέρουμε πολύ καλά. Χρειάζονται λοιπόν ε, τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τεχνολογία στη δασκαλία και περισσότερη υποστήριξη σε προσωποποιημένη διδασκαλία για ε, μαθητές με σε μειονεκτική θέση. Ωστόσο, το 80% των δασκάλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ιδιαίτερη σημασία αποδίδουν στο επάγγελμά τους, ε, το εκτιμούν ιδιαίτερα, το αγαπούν πολύ. Ωστόσο, μόνο το 20% βλέπει ότι η κοινωνία στην οποία ζουν έχει την ίδια εκτίμηση για το λειτουργήμα αυτό. Είναι δηλαδή ένα μοναχικό επάγγελμα και καθήκον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων είναι να εξασφαλίσουν δεν θα αισθάνονται τέτοια μοναξιά και τόσο βαρύ στους μοναχικούς τους ώμους το καθήκον της μετάδοσης της γνώσης στα παιδιά μας. Αυτό είναι νομίζω το θεματολογία για το μέλλον. Να εξασφαλίσουμε την καινοτομία, την αλλαγή, την ευελιξία στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και να στηρίξουμε το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Τι μπορούμε να κάνουμε. Μέσα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ένα είναι το Εράσμους και θέλω να υπογραμμίσω πως το Εράσμους δεν είναι απλώς ένα μέσο κινητικότητας των φοιτητών είναι μία από τι δυνατότητε, του, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να προσφέρει και δυνατότητε για αλλαγέ. εάν το χρησιμοποιήσουμε για να αξιοποιήσουμε και να υποστηρίξουμε την καινοτομία, τι καινοτόμε τάσει, τι ανταλλαγέ μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Έχει τεράστιο δυναμικό το εράσμου. Το έχουμε προετοιμάσει και σχεδιάσει μαζί με τα κράτη-μέλη, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί και στην ανάγκη για καινοτόμε αλλαγέ και προσαρμογή στη τεχνολογία. Έχουμε επίση και μέσα στο Εράσμου άλλα εργαλεία ή επιπλέον εργαλεία, το εκπαιδευτικό δίκτυο που αναφέρθηκε νωρίτερα. Έχουμε μια ε, πλατφόρμα ηλεκτρονική με 300.000 δασκάλους που εκπροσωπούν τεράστιο αριθμό σχολείων με ένα πάρα πολύ ισχυρό εργαλείο που μπορούμε και πρέπει να αξιοποιήσουμε περισσότερο και για να προαγάγουμε την τεχνολογία ως παιδαγωγικό εργαλείο και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε μέσω του Erasmus Plus για να υποστηρίξουμε τα, σχολεία είναι να προωθήσουμε την ηλεκτρονική αδελφοποίηση μέσα από μία πύλη ηλεκτρονική ε, σχολικής εκπαίδευσης. Schooleducation.eu είναι ο ψηφιακός της ιστότοπος και αυτό μπορεί να δώσει απαντήσεις για τον εκπαιδευτικό, για τον μαθητή, να αναζητεί τη γνώση και την ποιοτική προσέγγιση όπου βρίσκεται. Αυτό κάνουμε και ελπίζουμε το Κοινοβούλιο να μας υποστηρίξει και για να προαγάγουμε για το μέλλον το School Education Gateway, ώστε να καταστεί ένα πιο ε, στεναρό εργαλείο. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω και να προσθέσω ότι έχουμε προγράμματα για την καινοτομία στην εκπαίδευση. Η καινοτομία είναι γλώσσα, ε, λέξη του σειρμού. Πρέπει όμως να την εντάξουμε και στην εκπαίδευση. Και αυτό σχετίζεται, όπως ανέφερα και νωρίτερα, με τη συνεργατική εργασία και την διατομεϊκότητα, όπως είπα και νωρίτερα. Εάν θέλουμε τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, οι φοιτητέ και οι δάσκαλοι, οι μαθητές να ωφελούνται από τη νέα τεχνολογία, όπως θα πει και ο Ρομπέρτο, πρέπει να φροντίσουμε περισσότερες, να προσφέρουμε περισσότερες δυνατότητες τεχνολογικές στα σχολεία και πέραν των ε, επιστημονικών και τεχνολογικών ε, μαθημάτων, μαθηματικά φυσική και τεχνολογίες κλπ. Να προσφέρουμε και κατάρτιση στην, ε, στις τέχνες, στα καλλιτεχνικά δηλαδή τη μουσική και ούτω καθεξής. Θα πρέπει να έχουμε μαθητές οι οποίοι θα είναι ικανοί όχι μόνο σε ένα τομέα ανθρωπιστικές επιστήμες Φερρυπίν ή μόνο τεχνολογικές, αλλά σε όλες. Και μόνο έτσι μπορούμε να φέρουμε ουσιαστικές βελτιώσεις στον τρόπο με τον οποίο διδάσκονται και μαθαίνουν οι μαθητές. Αυτό είναι μια δυνατότητα που μπορεί να μα προσφέρει τεχνολογία και με βέβαιο ότι ο Ρομπέρτο θα προσθέσει σε αυτόν τον τομέα ακριβώ. Ευχαριστώ, λέει η κυρία Κώστα, και βεβαίω ε, μεγάλη είναι η πρόκληση και για μα στο πλαίσιο τη ευρωπαϊκή στρατηγική να ενταχθεί η καινοτομία με αυτόν τον ολιστικό τρόπο που αναφέρατε και να έχει πιο κεντρικό ρόλο η εκπαίδευση. Δίνω το λόγο στον κύριο Ρομπέρτο Βιόλα τώρα για την παρέμβασή του Σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πρόεδρε. Η DigiConnect θεωρεί ιδιαίτερη τιμή τη δυνατότητα που δίνεται να παραστεί σε αυτό το εργαστήριο. Νομίζουμε ότι αυτό σηματοδοτεί και μια μεγάλη πρόοδο στη συνεργασία μεταξύ των θεσμών για το πολύ σημαντικό αυτό θέμα και ο συνάδελφος ε, Χαβιέρ εστίασε ουσιαστικά στον πυρήνα του ζητήματος και μου άφησε την περιφέρεια, ε, το γύρω-γύρω, τέλος πάντων. Ε, και αυτά σημαντικά είναι. Χαίρομαι που είμαι ένας μειονοτικός μπλεκόσας, αλλά τέλος πάντων. Είμαστε και εμείς σημαντικοί, γιατί είναι σαφές ότι η τεχνολογία είναι ένα μέσο και έτσι πρέπει να παραμείνει. Είναι σαφές ότι η αλλαγή στα σχολεία παγορεύεται από τη μαθησιακή διαδικασία και όχι από την τεχνολογία. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας πάντοτε. Φανταστείτε όμως ένα σχολείο χωρίς ρεύμα ή χωρίς νερό. Είναι αυτό κάτι που μπορεί κανείς να το διανοηθεί στις μέρες μας. Νομίζω μπορεί κανείς να πει ότι ένα σπίτι χωρίς ε, σύνδεση μπορεί να θεωρηθεί κάτι αντίστοιχο με ένα σχολείο χωρίς νερό ή ρεύμα. Και στόχος μας τώρα είναι και οι αίθουσες δασκαλίας να συνδέονται στο διαδίκτυο, γιατί αυτό μπορεί ε, να βοηθήσει την προσαρμογή στο μεταβαλλόμενο κόσμο. Δεν είναι ένα ατού, είναι ένα ε, πλέον προαπαιτούμενο, είναι μια προϋπόθεση. Γι' αυτό και το θέμα των υποδομών έχει σημασία. Η σίγουρα είναι ένα μέσο, όπως είπα, και Χαίρομαι που είμαστε ένα μέρος εμείς, ε, σημαντικό όμως παρόλα αυτά, γιατί είναι πάλι επαναλαμβάνω σαν να μπορεί να υπάρξει ένα σχολείο χωρίς ρεύμα και χωρίς νερό. Όσο γάμα δελτα Connect, πολύ χαρά συνεργαζόμαστε από κοινού με τη γάμα δελτα ΕΑΚ και διαθέτουμε την πολιτική και του πόρου που έχουμε στη διάθεσή μα για την επίτευξη αυτού του στόχου, που είναι ένα από του σημαντικότερου στόχου για τι επικοινωνίε, αυτή η ελεύθερη εκπαίδευση δηλαδή. Υπάρχει συζήτηση, σημαντικό διάλογο και από αυτόν προκύπτουν συγκεκριμένε δράσει, μία από τι οποίε είναι κάθε αίθουσα δασκαλία να συνδεδεμένη στο διαδίκτυο και μάλιστα παρακολουθούμε την κατάσταση με τις τεχνολογίες πληροφορών και επικοινωνία στα σχολεία θα έχουμε κάποια αποτελέσματα και θα σας δώσουμε και τα σχετικά πορίσματα. Τώρα, η ε, σύνδεσιμότητα, δύο πτυχές έχουμε στα σχολεία να μπορούν να εκμεταλλευτούν ε, την αιχμή της τεχνολογίας και γι' αυτό τα σχολεία θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συνδέονται στις καλύτερες δυνατές τεχνολογίες. Οπτικές, ε, ίνες, υπερευριζωνικά δίκτυα κτλ. Έχουμε απλή, ε, διάφορες εφαρμογές, ε, ε, τα λοιπά. Και η διαδραστικότητα είναι σημαντικά πράγματα όλα αυτά. Η τεχνολογία, η δορυφορική τεχνολογία επίσης βοηθάει. Και όπως είπε και ο διευθυντής του Schoolnet, είναι σημαντικό και τα μικρά σχολεία να είναι το ίδιο καλά συνδεδεμένα με μεγάλα σχολεία. Αυτά που είναι στα κέντρα των πόλεων, για παράδειγμα. Γι' αυτό το είχαμε δει τα Connect ε, παρακολουθεί ε, ή ακολουθεί ένα διπλό δρόμο. Δηλαδή θέλουμε να βλέπουμε τι γίνεται με τη συνδεσιμότητα και την τεχνολογία στα σχολεία, αλλά θέλουμε όλα τα σχολεία να είναι συνδεδεμένα. Με την ΕΣΟΑ ε, δρομολογήσαμε αυτή την πύλη που την ανέφερε η Άρτη ε, για να είναι συνδεδεμένοι όλη η Ευρωπαϊκή πολίτες. Θέλουμε να προχωρήσουμε με την ΕΣΟΑ και με τους άλλους μας εταίρους, όσους θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτή την πρωτοβουλία, για να προωθήσουμε τα συνδεσιμότητα των σχολείων. Ως κάτι το οποίο μπορεί να ξεκινήσει μεν πιλωτικά, να καταστεί λειτουργικό σύστημα, αν θέλετε. Για το πιλωτικό πρόγραμμα φυσικά και θέλουμε να το υποστηρίξουμε, παρότι είναι περιορισμένοι οι πόροι μας, Σίγουρα μπορούμε όμως να συνεισφέρουμε. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τα λειτουργικά συστήματα, τα διαρθρωτικά ταμεία και τα κονδύλια που διέτρεψε στα κράτη-μέλη και το Ταμείο Επενδύσεων πρόσφατα ε, ακούσαμε ότι έχει και στόχο τη συνδεσιμότητα. Νομίζω ότι όλα αυτά τα κονδύλια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δημιουργήσουν ένα σταθερό σύστημα για τη διασύνδεση των σχολείων. Η συνδεσιμότητα λοιπόν, ναι, δεν είναι ο απότατο στόχο, αλλά είναι ένα βασικό βήμα. Το δεύτερο βήμα είναι η καινοτομία στην αίθουσα διδασκαλία. Χωρίς να το αποσυνδέσουμε αυτό βέβαια από το βασικό εκπαιδευτικό στόχο. Όπως ακούσαμε σήμερα, είναι σημαντικό να στηριχθούν οι διδάσκοντες, να υπάρχουν κατάλληλες πλατφόρμε για να μπορούν να πειραματίζονται οι δάσκαλοι να βιώνουν διαφορετικά ε, τη διδασκάλια και τη μάθηση. Τα τελευταία χρόνια η ΔΕΛΤΑ Connect υλοποίησε ένα πρόγραμμα και έχει επενδύσει 185 εκατομμύρια ευρώ στην έρευνα και την καινοτομία στη μάθηση μέσω τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών. Πρόσφατα είχαμε προκήρυξει και ένα διαγωνισμό που λέμε ότι 52 εκατομμύρια ευρώ θα τα διαθέσουμε σε τεχνολογίες για καλύτερες συνθήκες μάθησης και μιλάμε για πολλές τεχνολογίες, χρήση της εικονικής πραγματικότητας, τεχνολογίες παιγνίων, τεχνητή νοημοσύνη. Όλα αυτά τα χρησιμοποιούμε για να βελτιώσουμε τη μαθησιακή εμπειρία, για να έχουμε πραγματικά ένα σχολείο του μέλλοντος. Ουσιαστικά θέλουμε να, αν θέλετε, να μιμηθούμε την πραγματικότητα, να μπούμε σε μια πραγματικότητα που θα έχει και μια ψηφιακή διάσταση και ταυτόχρονα να κατανοήσουμε καλύτερα ε, τη μαθησιακή διαδικασία. Να στηρίξουμε τη συναισθηματική νοημοσύνη, το ανέφεραν οι δύο βασικοί ομιλητές. Η τεχνολογία πρέπει να βελτιώσει την βελτιωμένη αυτή ε, μαθησιακή εμπειρία του ανθρώπου Είμαστε ηγέτες ως Ευρώπη σε αυτήν την προσπάθεια και ελπίζω ότι μέσω της ε, υποστήριξης και από τη σχολική κοινότητα και με τα προγράμματα τα ερευνητικά που έχουμε μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο. Επίσης, ένας άλλος μας στόχος είναι να έχουμε ένα ψηφιακό μαθητή, φοιτητή, δηλαδή ένα μαθητή φοιτητή που θα είναι συνδεδεμένο σε αυτές τις υπηρεσίες, να έχει ηλεκτρονική ταυτότητα για να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτές τις νέες υπηρεσίες. Αυτό νομικά καθίσταται δυνατό με τη νέα με τον νέο κανονισμό περί ηλεκτρονικής υπογραφής που εγκρίθηκε πέρυσι από Κοινοβουλίο και Συμβούλιο. Λοιπόν, οι μαθητές, οι φοιτητές να είναι το πρώτο πείραμα εντό αγωγικών σε αυτή την ε, δυνατότητα διασύνδεσης. Επίσης, τα ψηφιακά, οι ψηφιακέ δεξιότητε θα πρέπει να εμπεριέχονται σε όλε τι πτυχέ σε κάθε γωνιά του σχολείου. Αλλά πρέπει να δούμε και τι συγκεκριμένε δεξιότητε απαιτούνται για να μπει κανεί σε αυτόν τον κόσμο των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνών και να μπορεί να εργαστεί σε αυτόν τον κόσμο. Ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας ICT υπάρχουν που δεν έχουν καλυφθεί και αυτό είναι παράδοξο λαμβανωμένο υπόψη στο μεγάλο ρυθμό ανέργων και, και νέων ανέργων, νεαρών ανέργων. Άρα μπορούμε να καλύψουμε αυτά τα κενά Γιατί αν αποκτήσουν ε, οι νέοι κυρίω, αλλά και άλλοι συνανθρωποί μα ψηφιακέ δεξιότητε, μπορούν να κλείσουν αυτά τα κενά, να καλυφθούν αυτέ οι θέσει εργασία. Τρει άξονε λοιπόν, στη συνδεσιμότητα, τεχνολογία, στην εκπαίδευση ψηφιακέ δεξιότητε. Η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Κονέξ σε αυτού του τρει άξονε θα συνεργαστεί με τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΕΑΚ στενά και με τι άλλε ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ, τι άλλε γενικέ διευθύνσει. Θα προωθήσουμε τη θεματολόγια αυτό και με τα χαρά βέβαια θα στηρίξουμε και το Κοινοβούλιο σε οποιαδήποτε δράση θέλησε να προωθήσει. Τους επόμενους μήνες τώρα αυτό το θεματολόγιο νομίζω ότι μπορεί να πλαισιωθεί από πολύ συγκεκριμένες δράσεις και ίσως τέτοιου είδους ακροάσεις αντισημερινή μπορούμε να ε, επαναλάβουμε και θα μπορούσαμε να εστιάσουμε σε μια προσεχή ευκαιρία σε ε, τρεις-τέσσερις βασικούς άξονες που θα θέλαμε να προωθήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ε, σας ευχαριστώ πολύ. Οι προτάσεις σας είναι πολύ σοβαρές και σωστές οι προοπτικές τις οποίες ανοίγουν οι δύο τελευταίες παρεμβάσεις, οι οποίες είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους. Το εκπαιδευτικό κομμάτι από τη μία, η δυνατότητα να ακολουθήσουμε τις γραμμές της αυξημένης συνδεσιμότητας, να καταστήσουμε όλες τις τάξεις και τα σχολεία συνδεδεμένα και το θέμα της καινοτομίας των σχολικών τάξεων. Χαιρετίζω εδώ τον καθηγητή Μπιόντι, αλλά τρίτο θέμα το οποίο υπογράμμισαν οι προλαλήσαντες είναι το θέμα των ψηφιακών ικανοτήτων σε σχέση και με τις προτάσεις τις οποίες αρχικά κάναμε της λεγόμενης ηλεκτρονικής ταυτότητας ή της e-κάρτας που έχει ζητήσει και το Φόρουμ του Ευρωπαϊκού είναι κάτι που ενδιαφέρει τους νέους και έχει μεγάλες πρόπτικες. Θα δώσω το λόγο τώρα στους συναδέλφους που έχουν ζητήσει το λόγο, με ταχύτητα όμως. Νομίζω ότι η συνάντηση αυτή ήταν ένα πρώτο βήμα, αν θέλετε, για την παρουσίαση της στρατηγικής για τον ψηφιακό χώρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το ρόλο που μπορεί να παίξει στον τομέα της εκπαίδευσης. Εμείς σαν Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας θα στηρίξουμε όσο μπορούμε την αναγνώριση αυτής της προτεραιότητας στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Σίλβια, ευχαριστώ πολύ τους ομιλητές μας. Σύντομη ερώτηση. Κυρίως προς τον κύριο Βιόλα, μιλάμε όχι μόνο για συνδεσιμότητα, δηλαδή όχι μόνο για τεχνολογικά ζητήματα, αλλά μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και το θέμα του περιεχομένου, content της εκπαίδευσης. Άρα τίθεται και το ζήτημα των Open Educational Resources, των, ανοιχτά, των δημόσια προσβάσιμων εκπαιδευτικών πόρων. Θέλω λοιπόν τη δική σας γνώμη για την ε, παραγωγή και διάθεση τέτοιων δημόσια προσβάσιμων εκπαιδευτικών πόρων. Υπάρχει κάτι σε σχέση με την ε, διάθεσή τους ελεύθερα στο κοινό, με την αδειοδότησή τους. Μπορεί κάτι να εμποδίσει την διάθεσή τους. Και έχω βέβαια υπόψη ε, το θέμα που θα μας απασχολήσει λίγο καιρό, το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων. Και θέλω να ρωτήσω σε ποιο βαθμό στον τομέα αυτό μπαίνουμε στα καλούπια του δικαίου, του πνευματικού δημιουργού και πόσο εύκολο ή δύσκολο μπορεί να γίνει για τον δάσκαλο να χρησιμοποιήσει ψηφιακό περιεχόμενο και πόσο θα κινδυνεύει ένας δάσκαλος μια δασκάλα με φυλάκιση αν προσφέρει γνώση από το ψηφιακό αυτό το περιεχόμενο στους μαθητές του. Πού βλέπετε λοιπόν ε, τις μεγαλύτερες προκλήσεις σε σχέση με τις δημόσια προσβάσεις εκπαιδευτικές, με τους εκπαιδευτικούς πόρους. Μόργανο και μετά θα δώσουμε το λόγο για απαντήσεις. Κύριος Μόργανο, ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμη αυτή η συνάντηση για το δεύτερο τμήμα. Έχω την εξή ερώτηση σε σχέση με τη δυνατότητα χρήσης των δυνατοτήτων που υπάρχουν και την ε, παραγωγή στις νέες τεχνολογίες, γιατί οι τεχνολογίες υπήρχαν πάντα, αλλά νέες τεχνολογίες τώρα είναι το θέμα μας, ψηφιακές δηλαδή πτυχές που απασχολούν τη συνάντησή μας και αν ε, μπορούν να προσφέρουν πραγματική υποστήριξη στην ουσιαστική και στην πραγματική δουλειά του εκπαιδευτικού. Η εμβάθυνση λοιπόν για τα πανεπιστήμια και η επιλογή της μη υιοθέτηση ή επιλογής της, ε, του ρόλου του εκπαιδευτικού στο πανεπιστήμιο, του καθηγητή, έχει να κάνει και με τις τεχνολογικές δυνατότητες που προσφέρονται. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε, να αναγνωρίσουν οι εκπαιδευτικοί ότι υπάρχει η αναγνώριση. Έστω και αν τώρα τη βλέπουν ως μία παρκή. Είναι, νομίζω, μία εικόνα άλλη αυτή που έχουμε όταν βγαίνουμε από το εκπαιδευτικό σύστημα και άλλη αυτή ε, όταν ε, μπαίνουμε σε αυτό. Γι' αυτό λοιπόν και μια προκλητική θα έλεγα ερώτηση θα έπρεπε, με βάση τα όσα ακούσαμε, τα θέματα αυτά να μην θεωρούνται στις συζητήσεις μεταξύ των κρατών ως δαπάνες, αλλά ως επενδύσεις. Αυτό το λέω ότι πρέπει να γίνει σχετική επιλογή. Πρώτα και μετά τις διατυπώσεις τις βρίσκουμε. Θα είναι η Ευρώπη αυτή που θα αναλάβει απευθείας ε, την διάθεση, θα είναι κάποιες επενδύσεις που θα μπορέσουν έμεσα να προσφέρουν τις δυνατότητες. Πάντως πρέπει πρώτα απ' όλα να εκφραστεί η βούληση για να αλλά αυτή φαίνεται να καθυστερεί ακόμη, να εκδηλωθεί. Και επίσης η συνάδελφος ε, Κάμερβερτ μίλησε στην ε, τοποθέτησή της για την δυνατότητα της πρακτικής αξιολόγησης, αξιοποίησης του περιεχομένου. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ευχαριστώ, Φερχέιβεν. Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο σημεία αυτά που είπε η κυρία Κάμερεβερτ καταρχάς για τις δυνατότητες σχετικές με την αδειοδότηση των, ε, του ε, προσβάσιμου υλικού και περιεχομένου και πώς το professional content, το, το ε, περιεχόμενο το οποίο βρίσκεται στη διάθεση των επαγγελματιών της ε, εκπαίδευσης μπορεί να περιγραφεί και να διατεθεί στους εκπαιδευτικούς. Αλλά βέβαια πάντοτε με επαλήθευση της ποιότητας. Ένα διδακτικό υλικό δηλαδή το οποίο δεν είναι ποιοτικό δεν μπορεί να βοηθήσει απαραίτητα. Υπόθηκε και νωρίτερα ότι πολλές φορές το διαδίκτυο μπορεί να εξυπηρετήσει την συλλογή πολυσχηδών πληροφοριών αλλά η ποιότητά τους δεν επαληθεύεται πάντοτε. Στον τομέα όμως της πρέπει πάντοτε να υπάρχει η ποιότητα. Αυτό και σε σχέση με τους οδηγούς σπουδών και σε σχέση με το εκπαιδευτικό υλικό που θα προσφέρει ο διδάσκων. Αυτό λοιπόν θέλω να κοιτάξουμε και επίσης, χωρίς μικρόφωνο, για τα δίκτυα των εκπαιδευτικών. Πολλοί ομιλητές μίλησαν και για τα δορυφορικά συστήματα και για την, ε, τις οπτικές σύνες ε, για την ευρυζωνική επικοινωνία. Υπάρχει η δυνατότητα της διασύνδεσης σχολείων, πανεπιστημίων, ανωτερών ιδρυμάτων με έναν τρόπο αξιόλογο, αξιόπιστο και λειτουργικό εξαρτάται αυτή η διασύνδεση, η συνδεσιμότητα καλύτερα από την υπηρεσία που θα προσφέρει η κάθε εταιρεία που έχει το ρόλο του παρόχου σε μια συγκεκριμένη περιοχή ή μπορούμε να έχουμε ισότιμο επίπεδο συνδεσιμότητας για όλη την Ευρώπη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ περιμένω τις απαντήσεις σύντομα, ανάλογα με το ποιο θεωρεί πως, το ε, τον αφορούν οι ερωτήσεις. Να ξεκινήσουμε από τον ε, τελευταίο, καθηγητής Βιόλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ίσως θα πρέπει να μιλήσω για την ελεύθερη εκπαίδευση, ανοιχτή εκπαίδευση και την πνευματική ιδιοκτησία. Δεν θα ήθελα να σας διαβάσω το κείμενο της ψηφιακής στρατηγικής, το οποίο θα δημοσιευθεί την Δετάρτη. Εμείς στην παρούσα φάση εξετάζουμε, λέει ο κ. Βιόλα, το συγκεκριμένο θέμα. Στα πλαίσια της διαβούλευσης, η εκπαιδευτική κοινότητα υπογράμμισε την ανάγκη υπογράμμισης των εξαιρέσεων και από την άλλη την προστασία του διδακτικού υλικού το οποίο ε, παράγεται και από ιδιωτικές επιχειρήσεις που είναι δραστήριες και στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Η Ευρώπη είναι ο πρώτος εξαγωγέας διδακτικού υλικού στον κόσμο. Δεν υπάρχουν απόλυτα, απόλυτη σύμπτωση συμφερόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας στο σύνολο της Ευρώπης ε, για την δυνατότητα χρήσης ελεύθερου διδακτικού υλικού και προστατευμένου από, πνευματικές, ε, από την έννοια της πνευματικής ιδιοκτησίας ε, εκπαιδευτικού υλικού. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν ένα ξεκάθαρο πλαίσιο για τις ε, επιτρεπόμενες ε, εξαιρέσεις, αποκλήσεις. Και θα συνεχίσουμε φυσικά την υποστήριξη της παραγωγής τέτοιου είδους υλικού εκπαιδευτικού υψηλής, ε, υψηλής ποιότητας, σημασίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει τα θέματα αυτά προσεκτικά και αναμένω αυτή τη στιγμή κατατεθεί η πρόταση να υποστηριχθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς θα σας βοηθήσουμε ως προς αυτό και η αδίποτε μορφή εμπλοκή σας ε, και συνεργασίας μαζί μας είναι επιθυμητή από πλευράς μας. Ε, λίγα λόγια για τις υποδομές επίσης. Νομίζω ότι η ουσία του πράγματος είναι να προσπαθήσουμε να βρούμε τον τρόπο ανάπτυξης της συνδεσιμότητας. Οι οπτικές ίνες δεν είναι παντού διαθέσιμες και γι' αυτό επιλέγουμε την βέλτιστη υποδομή όπου αυτό είναι δυνατόν. Και ταυτόχρονα επιλέγουμε μεγάλες πλατφόρμες για την σωστή εκμετάλλευση της συνδεσιμότητας. Άλλοι μπορεί να χρησιμοποιούν την οπτική ίνα, άλλοι μπορεί να χρησιμοποιούν το δορυφόρο, άλλοι το ψηφιακό σύννεφο. Ακολουθούνται διαφορετικά δίκτυα. Στόχος είναι ένα η συνδεσιμότητα. Και ο τρόπος επίτευξης του στόχου κάθε φορά ποικίλει. Για το θέμα το οικονομικό. Πράγματι το να λέει κανείς ότι η επένδυση στην εκπαίδευση δεν είναι κόστος, αλλά είναι πραγματική επένδυση. Α κοιτάξει κανείς χώρες όπως ε, η Δανία, η Ιαπωνία, βλέπουμε ότι οι Ιάπωνες πέτυχαν τα ίδια αποτελέσματα με τους Δανούς, αλλά με τα μισά χρήματα. Έχει σημασία λοιπόν να γνωρίζουμε ε, τι πηγαίνει καλά, τι πηγαίνει σωστά, τι σημαίνει εκπαίδευση και τι σημαίνει ουσιαστική εκπαίδευση. Η εκπαίδευση είναι ένας τομέας όπου είναι απαραίτητη η απόφαση, η λήψη πολιτικών αποφάσεων επί τη βάση συγκεκριμένων τεκμηρίων. Δεν είναι όμως πάρα πολύ συχνό αυτό. Πρέπει να δούμε τα θέματα της αποτελεσματικότητας και η εκπαιδευτική κοινότητα πρέπει να κάνει προσπάθεια εδώ. Δεν μπορεί από τη μία να πεσβεύει ότι οι δαπάνες για την εκπαίδευση είναι πολύ κρίσιμες και ταυτόχρονα να αρνείται την αξιολόγηση αυτής της δαπάνης. Ιδιαίτερα αν δει κανεί πόσο μεγάλη σημασία έχει η εκπαίδευση στα πλαίσια του ΑΕΠ των χωρών μελών. Λοιπόν, θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι τομείς οι φιλικοί προς τις επενδύσεις που οι χώρες μπορούν να δαπανίσουν χρήματα. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε και την εκπαίδευση και για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Και ταυτόχρονα να αναγνωρίσουμε ότι τα προβλήματα της εκπαίδευσης δεν εξαντλούνται στην χρηματοδότηση. Σε σχέση με αυτά τα οποία είπα, θα πρέπει να δούμε πώς συνδέεται η οικονομία με την εκπαίδευση. Βλέπουμε ότι ο υπόλοιπος κόσμος από την Αυστραλία στο Μεξικό, στην Ασία κτλ. δαπανούν περισσότερο τμήμα του ΑΕΠ τους από ότι μια μέση ευρωπαϊκή χώρα. Και αυτό πρέπει να μας κάνουν να σκεφτούμε για το αν η Ευρώπη δίνει επαρκή σημασία στην εκπαίδευση, στις δυνατότητες αλλαγής που μπορεί να προσφέρει η εκπαίδευση και κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει το μέλλον μας. Ευχαριστώ κύριε Διευθυντά. Ναι, και εγώ θα ήθελα πολύ σύντομα να μιλήσω για το ζήτημα των υποδομών που έθεσε η κυρία Φερχάη. Νομίζω ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους είναι τόσο πλούσια, αν θέλετε, η Ευρώπη είναι η ε, πολυμορφία της. Και αυτό ε, ισχύει και για τη γεωγραφική, ε, τη γεωλογική δομή. Υπάρχουν παιδινές, ορεινές τα λοιπά. Εάν η ουδετερότητα δικτύου γίνει εμπόδιο ουσιαστικά για την πρόσβαση ε, δεν θα ήταν κάτι θετικό. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες για να φτάσουμε σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους γιατί κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρίαση παραγωγική συζήτηση αυτό το απόγευμα και νομίζω ότι σε μια στιγμή στρατηγικής σημασίας τις παραμονές της παρουσίασης στρατηγική για το ψηφιακό ε, χάσμα, της Ευρωπαϊ... μέρισμα μάλλον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσδιορίσουμε προτεραιότητες και στρατηγικές για τις εκπαιδευτικές πολιτικές, για τις πολιτικές της καινοτομίας. Ε, προσπαθούμε και εδώ στο Κοινοβούλιο και την Επιτροπή μας να διατυπώνουμε σημαντικές εκθέσεις σε ζητήματα σχετικά με την πρόκληση αυτή και ιδιαίτερα βεβαίως διότι έχουμε πιστεύω όλοι μεγάλη ευθύνη να δώσουμε το πράσινο φως στη συνέχεια στις επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βάση προτεραιότητες αυτές και η συζήτηση που προκύπτει από τις δύο γενικές διευθύνσεις. Ευχαριστώ που ήρθατε ε, και εσείς. Ευχαριστώ πολύ για την ε, ε, πρόκληση που ήταν με την καλή έννοια η παρεμβάση των δύο πρώτων ομιλητών. Ευχαριστώ όλους τους άλλους ομιλητές. Νομίζω ότι διαπιστώνουμε πως η τεχνολογία δεν είναι μία συγκεκριμένη παρέμβαση ή ένας αυτός σκοπός για, ε, που πρέπει να ενσωματωθεί στην εκπαιδευτική στρατηγική, αλλά ξεκινώντας με τους διδάσκοντες ε, ένα εργαλείο για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το ίδιο ε, βοηθάει, όπως είπαμε με το Academy, με τα δίκτυα των σχολείων, πρωτοβουλίες που θα πρέπει βεβαίως να υποστηριχθούν και πρέπει να διαφυλαχθούν και στο βαθμό αυτονομίας που μπορούν να έχουν. Μπορεί λοιπόν σε αυτά η τεχνολογία να προσφέρει σημαντικές ε, συμβολές, σημαντική συμβολή για τα σχολεία, για τη δικτύωση, για την καινοτομία και στην οργάνωση του σχολικού περιβάλλοντος και βέβαια στο μεγάλο ζήτημα της συνδεσιμότητας που αναφέρθηκε νωρίτερα ως στρατηγικός στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε βεβαίως να δούμε συγκεκριμένες προτάσεις στα θέματα αυτά. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι ιδέες που ακούσαμε. Βεβαίως υπάρχει το ζήτημα της, του συσχετισμού μεταξύ της εκπαιδευτικής επένδυσης, της επένδυσης στην εκπαίδευση δηλαδή, με την αξιολόγηση της ποιότητας βεβαίως της της ε, επένδυσης, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να μιλήσουμε και για μια ελάχιστη ποιότητα, όχι μόνο ποσότητα επενδύσεων. Πρέπει λοιπόν από κοινού να δώσουμε το μήνυμα πως ξανακάνουμε επενδύσεις στο σχολείο, στην ε, εκπαίδευση, στον εκπαιδευτικό. Ώστε να είναι και για τον εκπαιδευτικό και για τις επόμενες γενναίες ε, θελκτικό το επάγγελμα αυτό και αυτό το λέω και προς την πρώτη ομιλήτρια, την καθηγήτρια από τη Φιλανδία, ότι η μεγάλη επένδυση για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών στη Φιλανδία ήταν εκείνη η οποία έδωσε αποτελέσματα ικανοποιητικά για τους ίδιους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν, αλλά ταυτόχρονα και ε, κατέστησε το λειτουργήμα του εκπαιδευτικού θελκτικό για τις επόμενες γενναίες. Αυτό είναι μια σημαντική προοπτική. Είναι επίσης πολύ σημαντικό το να έχουμε μέγιστες δυνατότητες ε, στη διάθεσή μας, δηλαδή και από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, για ε, άνοιγμα στην έννοια του πολίτη και για τον φοιτητή, να γίνει και ο φοιτητής ενεργός πολίτης, η δυνατότητα της ανάπτυξης αυτής της ευρωπαϊκής ταυτότητας του πολίτη και για τον φοιτητή, που θα διευκολύνει και η συνδεσιμότητα και το άνοιγμα στα μέσα και η δυνατότητα που θα καλύψει ακόμα και το κοινωνικό χάσμα, όπως αναφέρατε και εσείς μεταξύ των φοιτητών και εν τέλει βέβαια το πολύ λεπτό και ευαίσθητο θέμα που ανέφερε η κυρία Κάμερ Εύερτ της ε, προσβασιμότητας σε ε, προσβάσιμο, σε μη αδειοδοτούμενο περιεχόμενο για τους διδάσκοντες. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα λοιπόν η εμπειρία που έχω εγώ να σας περιγράψω από την ε, πατρίδα μου ιδιαίτερα όπου συμφώνησαν στην Ιταλία λοιπόν να, οι εκδοτικοί εκεί να δώσουν στα σχολικά ιδρύματα, στα, στις βιβλιοθήκες των σχολικών ιδρυμάτων, μια δυνατότητα πρόσβασης ελεύθερη. Νομίζω ότι με τέτοιες δυνατότητες, με τέτοιες πτυχές μπορούμε να παίξουμε για να κάνουμε πιο προσβάσιμη την ε, γνώση και ταυτόχρονα να ανοίξουμε μία αγορά, την αγορά των εκδόσεων στα σχολεία. Πάντα βέβαια με το σεβασμό των δικαιωμάτων των ε, ε, πνευματικών δημιουργών. Και το άλλο ζήτημα που έχει να κάνει με τη δυνατότητα που θα προσφέρεται στον ε, μαθητή, στο φοιτητή, να συνδέεται και να έχει συμμετοχική δραστηριοποίηση μέσα από ένα δίκτυο ε, στην εκπαίδευση. Για να καθίσετε η εκπαιδευτική διαδικασία πιο ενδιαφέρουσα. Αυτά λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όσα ακούσαμε. Και πριν κλείσει το θέμα αυτό και η συνεδρίασή μας, θα ήθελα να αναφέρω πολύ σύντομα κάτι το οποίο δεν είπα στην αρχή της συνεδρίωσης γιατί θέλω να ξεκινήσω την ακρόαση. Έχουμε τα τρία συνήθη θέματα της διαδικασίας μας, την έκρηση των πρακτικών δεν έχετε αντίρρηση. Το εγκύρι ράξος βέβαια της συνεδριάσεως που δεν έκαναν στην αρχή και την έκθεση για τα πεπραγμένα της αποστολής μας στην Ισπανία το Μάρτιο, που δεν θα μπορούσαμε να συζητήσουμε τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Τελειώνει εδώ η συνεδρία και συνεχίζουμε με τους συντονιστές και κλεισμένων των θυρών. Παρακαλώ λοιπόν, όποιος δεν έχει εργασία να αποχωρήσει από την αίθουσα.